βελτιωθούν ε, τα πράγματα ακόμα περισσότερο. Η ημερήσια διάταξη που έχουμε στα χέρια μας δεν προβλέπει αλλαγές, οπότε εγκρίνεται όπως έχει το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης. Ανακοινώσεις του ε, υποφαινομένου, τρεις στον αριθμό. Έχουμε εδώ συνεργείο τηλεόραση από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας του Κοινοβουλίου που είναι εδώ για να κάνουμε μια ταινία για τους επισκέπτες μας, πώς εργαζόμαστε, <laughs> προκενών εδράνων, εν πάση περιπτώσει, οι παρόντες πώς εργάζονται. Αυτό ήταν η πρώτη ανακοίνωση. Ανακοίνωση δεύτερη. Τώρα που συνεδριάζουμε εμείς στη Βόνη, στο Πέτερσπερκ συνεδριάζουν 45 υπουργοί ε, περιβάλλοντος από 45 κράτη και προσπαθούν και πάλι να δώσουν μια δυναμική στις διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή. Δυστυχώς τα πράγματα είναι ζωφερά από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία. Μάλλον έχουμε βάλει όπισθεν και θα πρέπει να φροντίσουμε να σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία. Και ίσως η συνάντηση στο Πέτερσπερκ να ε, αποβεί ωφέλιμη. Και στο μεταξύ έχουμε καταλήψει τη μεγάλη ιδέα της μεγάλης συμφωνίας και πάμε σε μικροσχέδια και μικροέργα. Δεν θα αρκέσει αυτό και ελπίζω για τον Ιούνιο για τη Βόνη, τη συνεδρίαση του ΟΗΕ θα έχουμε αιτήματα και πάλι να υποβάλουμε. Η τρίτη μου ανακοίνωση έχει να κάνει με τις πάρα πολλές ε, ψηφοφορίες που έχουμε αύριο για την έκθεση ε, IPPC και αυτά τα θέματα ξυλίας και τα νέα τρόφιμα. Είναι η κυρία Λιωτάρη, συγγήτρια για τα τρόφιμα, για το, την ξυλία η κυρία Λούκας και ο κύριος Κράμερ για το ε, IPCC. Κοίταξα τις τροπολογίες και μπορώ να σας πω προς χαρά της Επιτροπής να καταφύγω στο άρθρο 66 εδάφιο 3 που λέει εάν από την πρώτη μέχρι τη δεύτερη ανάγνωση μεσολαβήσουν ευρωεκλογές μπορεί ο Πρόεδρος να άρει τους περιορισμούς που κατά τα άλλα ισχύουν σε δεύτερη ανάγνωση και αναθεώρηση μια οδηγίας. Οπότε, για να μην αυθαιρετήσουμε, δηλαδή να, δεχτούμε κάποιες τροπολογίες επειδή αρέσουν στον ένα και να απορρίψουμε κάποιες άλλες επειδή αρέσουν στον άλλον, αποφάσισα να τις ε, εγκρίνουμε όλες, να είναι όλες ε, δεκτές. Θα ψηφίσουμε αύριο το πρωί να δούμε ποια είναι η πολιτική θέση ε, του νεοεκλεγμένου κοινοβουλίου για την παρούσα κοινοβουλευτική θητεία. Με μία εξαίρεση, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, στη δεύτερη ανάγνωση μπορούν να κάνουν τροπολογίες μόνο τα μέλη της Επιτροπής μας και ένα συνάδελφο ήταν πάρα πολύ επιμελής αλλά όχι μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Οπότε για το σημείο IPVC οι 124, 254, 205, 306 και 320 είναι μη παραδεκτές. Ο συνάδελφος Αντώνιο Ιντάλγο να με συμπαθάει, αλλά αυτά λέει ο οικονομισμό Πρέπει να είναι μέλος τη Επιτροπή Περιβάλλοντος. Πολιτικέ ομάδε λοιπόν να ε, προετοιμαστούν. Αύριο θα ψηφίσουμε όλε τι τροπολογίε. Τρία. Πρακτικά. 15-17 <laughs> Μαρτίου, αν δεν έχετε παρατηρήσεις. Εγκρίνουμε τα πρακτικά. Και πάμε στο σημείο 4 της ημέρης της διάταξης. Η γνωμοδότηση που ανέλαβα εγώ για μια έκθεση του συναδέλφου Σάιερ, άλλη μια έκθεση του συναδέλφου Σάιερ. Στη συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε αυτά τα δύο νέα άρθρα 290 της ε, ε, ανάθεσης ή χώρις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Νομοθετικών ε, Πράξεων. Κάναμε τη γνωμοδότησή μας στην πρώτη έκθεση του κυρίου Σάιερ και τώρα για το άρθρο 291 έχουμε τώρα πλέον τις εκτελεστικές ε, αρμοδιότητες και εδώ μας παρακάλεσαν να κάνουμε γνωμοδότηση. Τρία ε, πράγματα θα είχα να επισημάνω επί της ουσίας. Και πάλι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να είναι ισότιμοι και στη διαδικασία αυτή. Θα πρέπει να έχουμε εμείς όλη την πληροφόρηση που έχει και το Συμβούλιο ε, στη διάθεσή του. Ένα αυτό. Δεύτερο, σε θέματα περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας να μην υπάρχει κανένας περιορισμός γιατί η πρόταση έλεγε τη νέα διαδικασία, η διαδικασία αυτή η διαβούλευση ισχύει μόνο σε περίπτωση που το θεωρεί αυτό σκόπιμο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ έχω την εντύπωση και τη γνώμη ότι τα θέματα περιβάλλοντος και δημόσιας είναι πολύ ε, χρήσιμα και σημαντικά για τους πολίτες και αυτή η διαδικασία θα πρέπει να ακολουθείται σε όλα τα θέματα. Και το τρίτο είναι πιο τεχνικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θέλει όλες τις διαδικασίες μέχρι τώρα και τη ε, διαδικασία αυτή ε, κανονισμού να τις μεταφέρει στη νέα διαδικασία διαβούλευσης. Με την παλιά όμω διαδικασία εμεί έχουμε περισσότερε αρμόδιότητες και εξουσίες στο Κοινοβούλιο και αυτό προτείνω ε, να εξετάζεται αυτό ένα περίπτωση και όχι αυτόματα να μετατραπούν όλες οι παλιές διαδικασίες ή να καταργηθούν όλες οι παλιές διαδικασίες και να ισχύει μόνο καινούργια. Η κανονιστική διαδικασία, δηλαδή από την παλιά επιτροπολογία και τη σχετική απόφαση να διατηρηθεί. Αυτά για τη ουσία, τρει βελτιώσει που ε, προτείνω από πλευρά μα. Ο συνάδελφο Σάιερ, είπαμε, είναι εισηγητή και θα μα πει και αυτός τι θα κάνουμε τη δική μας γνωμοδότηση για την νομική επιτροπή και θα γνωμοδοτήσουν και άλλες επιτροπές για να πάει το θέμα στην Ολομέλεια. Παρατηρήσεις παρακαλώ. Κυρία Λεπάς. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση. Όχι σχετικά με αυτά τα οποία εσείς είπατε, αλλά αν κατάλαβα καλά και θα με διορθώσετε, για τη μεταφορά κάποιων αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου άμεσα στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και στην Επιτροπολογία για κάποια τεχνικά θέματα όπως ε, τα γενετικά τροποποιημένα και όχι μόνο. Υπάρχει ένας κίνδυνος εδώ. Ένας κίνδυνος ο οποίος θα καταστήσει ακόμα πιο δύσκολη την παρέμβασή μας στο μέλλον εφόσον όλα ρυθμίζονται σε επίπεδο επιτροπολογίας. Διορθώστε με αν δεν κατάλαβα καλά. Στην περίπτωση που κατάλαβα καλά, διαρωτώ με αν μπορούμε να κάνουμε κάποια διορθωτική πρόταση. Ε, εντάξει, υπάρχει ένα άρθρο στη συνθήκη της Λισαβόνας και έχει νόημα τα εφαρμοστικά μέτρα να τα αναλαμβάνει η εκτελεστική αρχή που είναι η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη αλλά η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει ότι το πλαίσιο για τη διαδικασία αυτών των εφαρμοστικών αρμοδιοτήτων θα αποφασίζεται από μας και από το Συμβούλιο. Οπότε μπορούμε τώρα να προσδιορίσουμε τα βασικά για τη διαδικασία που θα επιλογεί αργότερα με τα εφαρμοστικά μέτρα. Έτσι είναι σε κάθε κράτος. Η εκτελεστική εξουσία αναλαμβάνει την εκτέλεση εφαρμογή νόμων και το Κοινοβούλιο θέτει το γενικότερο πλαίσιο των ε, αρμοδιοτήτων εξουσιών της εκτελεστικής εξουσίας. Η Κομισιόν παρακαλώ να μας πει τη γνώμη της. Ο κύριος Αντουάν, όχι. Ε, εσείς είστε ο Μάριο Παύλο Τονρέρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ένα θα πω για το άρθρο 10 και την πρόταση της Κομισιόν για την αυτόματη, όπως λέμε, ευθυγράμμιση των παλιών διαδικασιών με τη νέα διαδικασία και τονίζω ότι η πρόθεση δεν είναι να αποκλείσουμε την ανάγκη ε, επαναξιολόγησης των παλιών κανονιστικών διαδικασιών που τώρα με τη νέα συνθήκη πρέπει να είναι κατα, κατεξουσιοδότηση πράξης. Αυτή η δουλειά πρέπει να γίνει παράλληλα με άλλο τρόπο. Οπότε το άρθρο 10 αυτό δεν το αποκλείει. Είναι μόνο μια τεχνική τροπολογία που θα αποφεύγει οι κανονιστικές ε, και διαχειριστικές επιτροπές που υπάρχουν θα συνεχίσουν να ισχύουν για πάντα, σύμφωνα με την απόφαση του 99, άμα δεν τα αλλάξουμε, και τότε θα έχουμε στο μέλλον ένα πολύ περίπλοκο ε, σύστημα με τις νέες διαδικασίες του κανονισμού και μετά θα έχουμε και τις διαχειριστικές και τις κανονιστικές διαδικασίες. Οπότε θέλουμε να τα πλουστεύσουμε όλα αυτά και ό,τι είναι διαχειριστικό και κανονιστικό σύμφωνα με την απόφαση του 99 θα είναι μια διαδικασία χωρίς να υπάρχει ανάγκη να επαναξιολογούνται οι πράξεις αυτές μετά και θα πρέπει να ενταχθούν στο άρθρο 290 για τις κατεξουσιοδότηση πράξης. Για τεχνικούς λόγους υπάρχει το άρθρο λοιπόν, χωρίς ε, να παραβλάπτονται οι άλλες διαδικασίες και τα άλλα θέματα. Ευχαριστώ για την παρατήρηση αυτή. Δεν ζητεί άλλο το λόγο. Αφού είναι μοιημένη φαίνεται. Βέβαια αυτό έχει μεγάλη σημασία για τη δουλειά μας. Λοιπόν, τα σημειώνω αυτά που είπαμε και η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι το μεσημέρι της 10ης Μαΐου, ενώ η ψηφο... Όχι, ναι, 10 Μαΐου το, στις 12 το μεσημέρι. Και πάμε τώρα στο επόμενο το οποίο είναι καθορισμός προτύπων για τις επιδόσεις των καινούριων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων όσον αφορά τις εκπομπές. Είναι ο Μάρτιν Κάλαχαν ο εισηγητής, ο οποίος ε, ε, ασχολήθηκε πολύ με το θέμα και θα μας το παρουσιάσει τώρα την έκθεσή του. Ορίστε κύριε Κάλαχαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε για την ευγενική σας εισαγωγή Χαίρομαι που φτάσαμε σε αυτό το στάδιο σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίου των ελαφρών εμπορικών οχημάτων. Ενθυμίστε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ουσιαστικά αντικατοπτρίζει κάποιες πλευρές της γενικότερης οδηγίας, του γενικότερου κανονισμού μάλλον για τις εκπομπές καυσαερίων που συζητήθηκε πέρυσι πριν την υιοθέτησή του αντικατοπτρίζει την πρόταση αυτή και σε σχέση με τους στόχους, με την οικοκαινοτομία, τις κυρώσεις κτλ. Νομίζω όμως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναγνώρισε ότι τα βαν αυτά, τα ελαφρά εμπορικά οχήματα, είναι αρκετά σημαντικά και ποσοστιαία εννοώ Άλλωστε πάρα πολλοί χρήστες οι οποίοι παρασύρθηκαν από το μάρκετινγκ και τις διαφημίσεις αγόρασαν μεγαλύτερα οχήματα από όσα χρειαζόντουσαν και <clears throat> δεν πιέστηκαν οι κατασκευαστές να παράγουν πιο οικονομικά εν πάση περιπτώσει οχήματα και αυτό ε, διευκόλυνε βέβαια και την κυκλοφορία οχημάτων τα οποία επιτρέπουν μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών. Βέβαια υπάρχει εδώ το θέμα της ε, χρηστικότητας των οχημάτων αυτών. Πολλές φορές είναι αρκετά γυμνά τα οχήματα αυτά, δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες μείωσης του βάρους. Και φυσικά το πιο αποτελεσματικό βάν είναι αυτό το οποίο έχει το σωστό μέγεθος θα έλεγα για το βάρος το οποίο μεταφέρει και ναι, φυσικά όταν κάποια εταιρεία χρησιμοποιεί δύο μικρότερα βαν για να μεταφέρει τα προϊόντα της, αυτό μολύνει περισσότερο. Έτσι λοιπόν το 90% των οχημάτων αυτών ε, είναι πετρελαιοκίνητα, κάτι το οποίο επιτρέπει στην εταιρεία, στις εταιρείες κατασκευαστικές να πετυχαίνουν στόχους κατανάλωσης. Σχετικά με τους υπόλοιπους στόχους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή <clears throat> έχει προτείνει ε, σταδιακή εισαγωγή των 175 γραμμαρίων το 2018 και μια μείωση 10 γραμμαρίων κατέτος ανάμεσα στο 2016 και το 2020 για να πετύχουμε το 2020 το 135 ε, γραμμάρια, κάτι το οποίο είναι πολύ πιο θα έλεγα φιλόδοξο από ότι το αντίστοιχο που προβλέπεται για τα επιβατικά οχήματα. Στην ουσία από το 2015 μέχρι το 2020 προβλέπεται μία μείωση 7 γραμμαρίων κατέτος, συνολικά δηλαδή 35 γραμμαρίων, κάτι το οποίο σαν μείωση συνιστά μία πάρα πολύ φιλόδοξη πρόθεση σε σχέση με τα αυτοκίνητα, τα οχήματα, τα ιδιωτικά. Εγώ προτείνω μία ελαφρά χαλάρωση να φτάσουμε στο 150 το 2020 το οποίο εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ φιλόδοξο, τεχνολογικά αντιπροσωπεύει μια σημαντική πρόκληση, αλλά είναι σίγουρα και πιο πραγματιστικό και έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, διατηρώντας φυσικά τους λόγους ύπαρξης του βαν, του εμπορικού αυτού οχήματος. Προτείνω επίσης περιορισμένες περιοριστές ταχύτητας, οι λεγόμενοι κόφτες ε, να ε, εισαχθούν σύμφωνα με, τις, ε, με τα στοιχεία τα οποία έχουμε υπάρχει αυτός ο μύθος ότι όπως τον περιγράφουμε στις Ηνωμένε Πολιτείες δηλαδή το, το εμπορικό όχημα φάντασμα συνήθως είναι λεφτά τα οποία κολλάνε στα πίσω φώτα σας στον αυτοκινητόδρομο και δημιουργούν ατυχήματα, προκαλούν ατυχήματα και δημιουργούν φοβίες Σχετικά τώρα με τις κυρώσεις, προβλέπεται όπως και για τα αυτοκίνητα 195 μάλλον γραμμάρι, ε, euro αναγραμμάριο, κάτι το οποίο είναι θα έλεγα σαν κύρωση ιδιαίτερα υψηλή. Προτείνω επίσης και σε σχέση με το συνδυασμό ε, των αυτοκινήτων αυτών τη συνδυασμένη χρήση. Κάποια από αυτά τα μοντέλα πολλές φορές ε, συνδυάζουν τον επιβατηγό ρόλο και τον ε, εμπορικό ρόλο, τον ρόλο μεταφοράς. Αυτό είναι λίγο στρεβλό το να πει κανείς ότι πρέπει να υπάρχουν δύο διαφορετικοί κανονισμοί ε, για ε, τα οχήματα αυτά και θα μπορούσαμε ίσως να πετύχουμε και διαφορετικές μορφές εξοικονόμησης εκπομπών εννοώ και θα πρέπει αυτόματα οι εκπομπές αυτές να ισχύσουν και για τα δύο είδη των οχημάτων και σίγουρα οι εταιρείε, ακόμα και όταν έχουν δύο διαφορετικές μονάδες παραγωγής των εμπορικών οχημάτων και των επιβατηγών οχημάτων, πρέπει να είναι σε θέση να συνδυάζουν την παραγωγή και να περνούν τα πλεονεκτήματα του ενός στο άλλο. Ένα ειδικότερο πρόβλημα είναι τα λεγόμενα πολυφασικά σε εισαγωγικά οχήματα. Ίσως να μην τα γνωρίζετε όσοι δεν ξέρετε καλά τον κανονισμό αυτό. Είναι οχήματα τα οποία πολλούνται ατελεί Δηλαδή οι πολίτες σαν παράδειγμα μόνο το αμάξωμά τους και η καμπίνα από τον κατασκευαστή και συνήθως δίδονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες προσθέτουν εκατοντάδες διαφορετικά τελειώματα, γερανούς, πλατφόρμες, ε, τροχόσπιτα, ό,τι θέλετε πάνω στο αμάξωμα αυτό. Αυτό δημιουργεί προβλήματα σε σχέση με την οδηγία πλαίσιο, με τον κανονισμό πλαίσιο, συγγνώμη, γιατί είναι πάρα πολλοί κατασκευαστές σε όλη την Ευρώπη, είναι μικροί κατασκευαστές και δεν είναι πάντα δυνατό να εφαρμοστεί σωστά ο κανονισμός για αυτούς, γιατί πετυχαίνουν τις εξαιρέσεις λόγω μικρού όγκου παραγωγής. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό εδώ ο αρχικός κατασκευαστής να είναι υπεύθυνο σύμφωνα με τον κανονισμό για το προϊόν αυτό. Οι κατασκευαστές βέβαια λένε ότι δεν είναι υπεύθυνοι για το σώμα το οποίο προστίθεται πάνω στο αμάξωμα. Νομίζω ότι η σωστή λύση και όχι αυτή την οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έλεγε ότι θα πρέπει να δοθούν ε, εικονικοί αριθμοί που θα πρέπει να γίνουν σεβαστοί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω ότι θα πρέπει να βρει ένα σύστημα να διαμορφώσει μια τέτοια διαδικασία έγκρισης τύπου σαν παράδειγμα έτσι ώστε ε, τα αυτοκίνητα αυτά να, να καταμετρώνται και να αξιολογούνται τη στιγμή όπου έχει τελειώσει η διαδικασία τους και είναι έτοιμα για κυκλοφορία. Εγώ δεν λέω ότι κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ εύκολο και θα πρέπει να δημιουργηθούν νέα συστήματα παρακολούθησης. Η παρακολούθηση θα πρέπει να είναι πάρα πολύ εντατική και πάρα πολλές φορές θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι οι κατασκευαστές δεν γνωρίζουν μερικές φορές ποια θα είναι η τελική κατάληξη των οχημάτων αυτών και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν να έχει ένα σύστημα παρακολούθησης της ολοκλήρωσης των οχημάτων αυτών και ε, αυτό να φαίνεται στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης τύπου. Αυτές είναι οι βασικές βελτιώσεις τις οποίες προτείνω για την πρόταση που μας έκανε η Επιτροπή. Θα περιμένω με ενδιαφέρον αυτά τα οποία θα πούνε και οι συνάδελφοι από τις ε, άλλες επιτροπές και τα μέλη φυσικά της επιτροπής μας. Ευχαριστούμε πολύ Μάρτιν Κάλλαναν για την έκθεση και την εργασία που έχετε κάνει μέχρι τώρα για να γίνει κάτω κατανοητός ο ειδικό αυτός τομέας των ελαφρών εμπορικών οχημάτων. Έχουμε εμπειρία ήδη ε, από τον περιορισμό εκπομπών ε, οχημάτων οπότε ε, είχαμε κάνει την αρχή η Άνια Βάις Γκέρμπερ ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή Μάρτιν Κάλλαναν για την πολύ ωραία έκθεση θεωρώ είναι πολύ επιτυχημένη γενικά και χαίρομαι για τη συνεργασία στη... είχαμε παρόμοια ε, αποτελέσματα και πολύ καλά και για τον περιορισμό εκπομπών άλλων κατηγοριών με επικοδομητική συνεργασία. Γι' αυτό είναι ε, προσβλέπω στη συνεργασία. Τώρα στις λεπτομέρειες, γενικά το σχέδιο είναι επιτυχημένο, αργότερα θα επισέλθω και στα θέματα που με βρίσκουν σύμφωνοι 100%. Νομίζω όμως ότι θα έπρεπε να είμαστε πιο ε, φιλόδοξη σε ό,τι αφορά τις οικοκαινοτομίες. Ο στόχος θεωρώ ότι πρέπει να είναι όχι τιμωρητικός μέσα από πρόστιμα ε, κάτι αντίστοιχο με τα φορτηγά, αλλά να δώσουμε περισσότερα κίνητρα ώστε να βγουν στην αγορά μηδενικής εκπομπής οχήματα ή τέλος πάντων με πολύ περιορισμένη εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Στις οικοκαινοτομίες και στα super credits μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Για το πρώτο θέμα των οικοκαινοτομιών είναι σημαντικό και στα βιοταχή να έχουμε ε, μείωση της γραφειοκρατίας μέσα από τις εφαρμοστικές διατάξεις ώστε να μπορέσει να κάνει ε, η βιομηχανία τέτοιες καινοτομίες αλλιώς δεν θα προχωρήσει. Με τον κύριο Όμνο από την Κομισιόν έχουμε μια συνάντηση ε, τώρα αυτή τη βδομάδα που ελπίζω ότι θα βοηθήσει και νομίζω ότι θα διαμορφώσουμε κάτι παρόμοιο στα ελαφρά εμπορικά. Ο περιορισμός στα 7 γραμμάρια μπορεί να συζητηθεί και πάλι, πάντως γενικά χρειάζονται κίνητρα σε αυτό το τομέα. Επίσης κίνητρα μπορούν να υπάρχουν και με τα super credits όπως τα λέμε, όπου ανταμείβονται οι κατασκευαστές που κατασκευάζουν οχήματα μηδενικής εκπομπής ή οχήματα που έχουν εκπομπή κάτω από 50 γραμμάρια. Η αναγνώριση όμως περιορίζεται μέχρι το 2016 και μάλλον μέχρι το 2016 θα είναι πολύ δύσκολο να υπάρχουν αυτοκίνητα σημαντικά σε αριθμό τα οποία θα κατέβουν κάτω από τα 50 γραμμάρια. Γιατί δεν κάνουμε ένα πιο μακρινότερο ορίζοντα ούτως και εγώ θα ε, υποβάλω σχετικές τροπολογίες και Συζήτησα και με τη συνάδελφη που ήταν ανοιχτή πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτά ήθελα να σας πω. Κατά τα άλλα συμφωνώ και με τον μακροπρόθεσμο στόχο με τον εισηγητή. 435, ε, 135 ε, ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ψηλός στόχος στις μελέτες της Κομισιόν και οι δαπάνες είναι 350 σε 125, 900. Ε, δεν υπάρχει μελέτη επιπτώσεων, τι θα σήμαινε δηλαδή αυτό. Απλώς κάποια στοιχεία δίνει η Κομισιόν και χρησιμοποιεί σε στόχο σε ε, γραμμάρια υψηλότερο. Αν είναι 7 με 9.000 ευρώ σε ένα κάντι, ας πούμε, το οποίο σε σχέση με την τιμή του και από οικονομικής και από τεχνικής άποψης δεν είναι εφικτός ο στόχος και για τον βραχυπρόθεσμο στόχο μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα. Μένουν οι στόχοι της Κομισιόν ε, και ε, όταν είναι ε, πιο μακροπρόθεσμο το πρόγραμμα θα μπορούσαμε να μείνουμε στους βραχυπρόθεσμους στόχους εκεί αλλά μακροπρόθεσμα χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Νομίζω ότι έχουμε μια συνεχή υποχρέωση, ένα phase-in μεταξύ βράχη και μακροπρόθεσμων στόχων να έχουμε συνεχή μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα ούτως ώστε να αναλάβουν μια μόνιμη υποχρέωση και οι βιομηχανίες, οι κατασκευαστές που θα πρέπει να ε, εργάζονται και με υποχρεωτικούς ενδιάμεσους στόχους. Νομίζω ένα τέτοιο συνεχιζόμενο phasing θα ε, επέτρεπε καλύτερο προγραμματισμό στη βιομηχανία και θα υποβάλω μια σχετική πρόταση. Ε, παρόμοια είπε και η Επιτροπή Βιομηχανίας. Τώρα για τον περιορισμό της ταχύτητας έχουμε τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Ε, εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Ούτε έχω δει μελέτη μέχρι τώρα που να ε, αποδεικνύει την εξοικονόμηση σε εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι τα αυτοκίνητα αυτά χρειάζονται κάποια απόδοση του κινητήρα ούτω ώστε να μπορούν να μεταφέρουν και το βάρος που ε, πρέπει να ε, μεταφέρουν. Έχει συσχέτιση αυτό με την ταχύτητα. Ε, στην τροπολογία, στην αιτιολόγηση γράφει ότι ο εισηγητής ότι δεν θα υπάρξει προηγούμενο. Θα δημιουργηθεί όμως προηγούμενο όταν εμείς έχουμε τόσο χαμηλή μείωση της ταχύτητας. Επίσης πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ανταγωνισμός με τα ιδιοταχή. 95 ευρώ αποφασίστηκε και τι όχι περισσότερο. Τώρα στα multi αυτά στα πολυφασικά νομίζω ότι η πρόταση του εισηγητή είναι επίσης καλός και μπορώ να συμφωνήσω γιατί για πολλοί κατασκευαστές ε, δεν ξέρουν ακριβώς τι ε, εξαρτήματα θα προσθεθούν στο βασικό όχημα. Δεν υπάρχουν δεδομένα, χρειάζεται συμβαστική πρόταση εδώ. Και τέλος το pooling, εδώ το βλέπουμε πιο, κάπως επικριτικά. Γιατί υπάρχουν βιομηχανίε που δεν δραστηριοποιούνται και στα γεωταχή και στα ε, επαγγελματικά. Οπότε ε, ε, αυτοί θα αδικηθούν. Πάντως νομίζω ότι θα βρεθεί μια καλή συμβαστική λύση και ευχαριστώ άλλη μια φορά για το καλό σας ε, σχέδιο έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βάισμπεργκερ. Ο Ματίας Κότεσε. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Μάρτιν Κάλαναν για την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά πρέπει να πω τότε ε, ήταν η έκθεση ακόμη για τα ΙΟΤΑΧΗ. Ε, τα ίδια συζητούσαμε ε, για αναβολή προθεσμιών, ημερομηνιών, για αποδυνάμωση και δεν είναι βελτίωση για τις οριακές ε, τιμές ε, ούτε η έκθεση Κάλαναν. Εκεί που ένιωσα ευχάριστη έκπληση και χάρηκα ήταν για το περιορισμό του ορίου ταχύτητας. Και σε σχέση με το όσα είπε η κυρία ε, Βάις Κέρμπερ, δεν θέλουμε να αλλάξουν τίποτα στον κινητήρα, αλλά να βάλουμε ηλεκτρονικό περιοριστή, κόφτη ταχύτητας. Να αποφασίσουν όμως οι κατασκευαστές οι ίδιοι τι κινητήρες θα φτιάξουν, τι δουλειά έχει να ανακατευθεί η πολιτική στην τεχνολογία των κινητήρων ε, ε, ο κάθε κατασκευαστή αποφασίζει πώς θα σχεδιάσει το κινητήρα του και εμεί καλά θα κάνουμε να μην τα αγγίζουμε αυτά τα πράγματα. Αλλά για τους κόφτες εντάξει, έχει νόημα. Διότι η αντίσταση του αέρα αυξάνεται ε, και τετραγωνίζεται στο τετράγωνο, ναι. Ε, και αυτό έχει επιπτώσει στην κατανάλωση των καυσίμων και στο κόστος. Λοιπόν, ναι στα μέτρα που ε, είναι αποδοτικά για το κόστος, που περιορίζουν το κόστος. Ναι για τον περιοριστή της ταχύτητας και γι' αυτό να υπάρξει επιβράβευση των κατασκευαστών που βάζουν τους κόφτες. Δηλαδή, αναγραμμάριο διοξιδίου ε, του άνθρακα να τους υπολογίζεται αυτό και να επιβραβεύεται και εδώ χρειάζεται σαφής ορισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πώς μπορεί να γίνει τεχνικά. Και όπως σας είπα, ευχαριστώ και ευγνωμονώ τον Μάρτιν Κάλλεν που ε, συμπεριέλαβε την ιδέα αυτή και στην Επιτροπή ε, Μεταφορών. διάφορες πολιτικές ομάδες το έχουν υιοθετήσει και εδώ πραγματικά μπορούμε να περιορίσουμε το κόστος και το διοξίδιο του άνθρακα στην πραγματική ζωή. Σε ό,τι αφορά την νομοθεσία ασφαλεία, ε, έχει και αυτό συνοδευτικέ ε, θετικέ επιπτώσει, αλλά αυτό δεν μα αφορά. Εμεί είμαστε Επιτροπή Περιβάλλοντο εδώ και αυτό θα πρέπει να εξετάζουμε και να ε, νομοθετούμε για το περιβάλλον. Τώρα, πιο μακροπρόθεσμα. 135 γραμμάριο στόχος είναι φιλόδοξος, αλλά χρειάζεται αλλαγή τεχνολογίας, διαφορετικές τεχνολογίες τα οχήματα, αλλά μας λένε όλοι οι οργανισμοί, Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, ότι μειώνεται το πετρέλαιο και αγωνιζόμαστε να βρούμε ε, πρώτες και αυξάνεται ο πληθυσμός της γης ταυτόχρονα. Γι' αυτό έχει νόημα να ε, βάζουμε κάποια όρια και στο δεξίδιο του άνθρακα και στα καυσαέρια και στα καύσιμα. Και είναι η βασική ιδέα αυτή της ε, πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό που μας ενδιαφέρει και στις νέες επενδύσεις είναι να περιορίζεται η κατανάλωση καυσίμων και να υπάρχουν νέα όρια. Αυτά είναι τα μακροπρόθεσμα. Τώρα, τα βραχυπρόθεσμα μέτρα και το, η προοδευτική εισαγωγή του, το phasing in. Πρέπει να σας πω ότι θέλω να συμφωνήσω με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πολύ ρεαλιστική και τα 175 γραμμάρια με σημερινέ τεχνολογίε που ήδη ε, υπάρχουν μπορεί να επιτευχθεί ο στόχο αυτό. 175 γραμμάρια. Αυτό να παραμείνει. Και ε, για το χρονοδιάγραμμα συμφωνώ επίση με την Κομισιόν. Ο στόχο του ε, εισηγητή δεν με βρίσκει σύμφωνα 140 γραμμάρια και μάλιστα από το 2025 είμαστε σε λάθος δρόμο, είναι κακό μήνυμα αυτό και από πλευράς οικονομικής, όχι μόνο τεχνολογικής είναι η βιομηχανία κλειδί η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και δεν την εξυπηρετούμε έτσι. Έχει τα καλύτερα προϊόντα στην αγορά και σε παγκόσμια αγορά. Και μόνο έτσι θα μπορέσει να ορθοποδήσει και να παραμείνει. Λοιπόν, έχουμε την κείμενη ε, νομοθεσία του 2008 για τα και Υπάρχουν μοντέλα τώρα και τύποι αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην αγορά. και στα 20 γραμμάρια ήμασταν σε ό,τι αφορά τον περιορισμό ε, των καυσαερίων και δυσκολεύεται πραγματικά η ε, βιομηχανία. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να το καταφέρει, αλλά μπορεί να το πετύχει αυτό το στόχο, πιστεύω. Και από πλευρά βιομηχανική πολιτική έχει νόημα. Για τα πρόστιμα τώρα. Συμφωνώ με τον ε, Γκάλανα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να είναι διαφορετικά τα πρόστιμα στα γεωταχή και στα ελαφρά δημόσια χρήση επαγγελματικά αφού είναι παρόμοια. Δεν έχει νόημα να έχουμε διαφορετικά μέτρα και σταθμά. 95 ε, ευρώ για τον ένα και 120 για τον άλλον. Αφήστε δε που δεν πιστεύω ότι θα πληρώσει κανένα κατασκευαστή. Συμφωνώ με τον εισηγητή. Για τα πολυφασικά, multi-stage, είναι πρόβλημα αυτό μεγάλη διαφορά από τα ιδιωτική χρήση και θα πρέπει να αναλάβουν τι ευθύνε του οι κατασκευαστέ, γιατί δεν ξέρουν τελικά τι θα γίνει με τα οχήματα αυτά. Γι' αυτό θεωρώ καλή και την πρόταση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λίγο να μα εξηγήσει τι θέλει να κάνει και πώ θέλει να προχωρήσει σε αυτό το σημείο. Συνοψίζω και συμπεραίνω. Είναι σημαντική η νομοθεσία αυτή. Δεν απέχουμε τόσο πολύ στο θέμα αυτό, ούτε είναι τόσο επίμαχο όπω η έκθεση Σακώνη θα συμφωνήσουμε πιστεύω, αλλά το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θα πρέπει να το αποδυναμώσουμε στις βασικές γραμμές, όπως κάνει ο Μάτριν που Αυξάνει τις οριακές τιμές και δεν ξέρω και αν είναι εφικτά αυτά, να τα ξανακοιτάξουμε τα πολύ φασικά και τα υπόλοιπα. Και θα χαιρόμουν να έχουμε περιορισμό ταχύτητα στην πράξη για περιορισμό και των καυσαερίων και της εκπομπής του διοξιδίου του άνθρακα με υπολογισμό πολύ σημαντικό όμως περιορισμό της ταχύτητας αλλά με μετρήσιμα μεγέθη. Και ε, περιμένω με ανυπομονησία τη συζήτηση και τη συνέχεια που θα δεθεί στο θέμα αυτό. Έχουμε συνολική ευθύνη αυτή τη στιγμή τα τάπα λέει ο πρόεδρος ότι συνεδριάζουν οι υπουργοί ε, περιβάλλοντος. Εντάξει. Ε, θα πρέπει να δείξουμε ότι μας ενδιαφέρει σοβαρά η προστασία του περιβάλλοντος από την κλιματική αλλαγή. Και να έχουμε και μια ευφυή βιομηχανική πολιτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η Όλγα Κράμερα για του φιλελευθέρου ή ο Κρι Ντέιβι. Ο Ευχαριστώ. Πολύ λυπάμαι που έγινε η εισαγωγή της νομοθεσίας έτσι σχετικά με τις εκπομπές του οξυδίου του άνθρακα. Ε, δεν είναι ήδη πολυτελείας αυτά τα οχήματα. Πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η αύξηση της απόδοσης των καυσίμων. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό μειώνοντας και τις εκπομπές. Ε, για τα και, τη νομοθεσία για τα καινούρια αυτοκίνητα υπάρχει μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση στο λόμπι του κλάδου. Ε, για πολύ καιρό δεν έχει υπήρξε καθόλου μείωση ούτε ε, του διοξείδιο του άνθρακα ούτε αύξηση της απόδοσης καυσίμων και τέλος υπάρχουν οι ε, προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου. Και τώρα έχουμε ξαφνικά μεγάλη μείωση του CO2. Και είπε μάλιστα η κυβέρνησή μας ότι αυτή ήταν η μεγαλύτερη μείωση που επιτέχθηκε τον τελευταίο καιρό και έγινε το ίδιο και σε άλλες χώρες. Από το 2001 μέχρι το 2007 η απόδοση καυσίμων των φορτηγών μειώθηκε γιατί οι κινητήρε ε, ήταν πιο ισχυροί. Αυτό που θα έλεγα λοιπόν για τι προτάσει του Μάρτιν Κάλαναν αυτό που με βρίσκει σύμφωνο είναι οι κόφτες, γιατί έτσι οι κατασκευαστές θα σχεδιάζουν τους κατάλληλους κινητήρες και όχι υπερβολικά ισχυρούς. Αυτό που υποτίμησε ο Μάρτιν είναι ότι αυτό, αυτή η βελτίωση στην απόδοση καυσίμων που θα προκύψει ως αποτέλεσμα πρέπει να λυθεί υπόψη γιατί είναι πιο εύκολο οι κατασκευαστές να ε, εξασφαλίζουν αυτές τις βελτιώσεις και παράλληλα να μειώνουν και το CO2 εκπομπέ. Τώρα, για τα αγιοταχή, η νομοθεσία είναι, δείχνει ότι η φιλόδοξη και σταθερή ε, νομοθεσία έχει αποτελέσματα. Η τεχνολογία, όπως αναφέρθηκε, η τεχνολογία υπάρχει. Ε, δηλαδή, οι κατασκευαστές, οι Γερμανοί συνήθως των εξαρτημάτων των αυτοκινήτων λένε ότι εύκολα μπορούμε να φτάσουμε τους στόχους αυτούς και μπορούμε να πάμε και στα 160 γραμμάρια ε, δηλαδή λένε, ας πούμε, δώστε μας την παραγγελία εσείς και εμείς θα τα καταφέρουμε. Θέλουν να πουλήσουν. Ε, είναι αυτοί οι συναρμολογητές που θέλουν να αναβάλουν τις αποφάσεις. Η τεχνολογία όμως υπάρχει. Ε, έχει δίκαιο ο προηγούμενος ομιλητής. Η Κομισιόν λέει ότι αν πούμε 135 γραμμάρια ως στόχο ε, διοξιδίου μέχρι το 2020 Κατά τη διάρκεια ζωής ο οδηγός θα εξοικονομήσει ένα ποσό σε ευρώ, 70 δολάρια το βαρέλι. Αυτά θα είναι οχήματα του 2020 που θα είναι στο δρόμο και το 2030. Δηλαδή θα είναι 70 δολάρια το βαρέλι, το 2030 το πετρέλαιο η εξοικονόμηση ενδεχομένως ε, από τα αυτοκίνητα αυτά είναι πολύ μεγαλύτερη τάξη μεγέθους από ό,τι στους υπολογισμούς που μας έκαναν γιατί οι τιμές του πετρελαίου θα είναι πολύ πιο πάνω. Βλέποντας λοιπόν τις προτάσεις του Μάρτιν Κάλαναν λέω ότι ε, προκρίνει κατασκευαστές ε, που είναι λιγότερο ικανοί. Υπάρχουν πολλοί που έχουν δώσει, έχουν κατασκευάσει αυτοκίνητα πιο οικονομικά από ό,τι εκείνα των ανταγωνιστών με μικρότερες ε, εκπομπές. Υπάρχουν παραδείγματα ορθής πρακτικής. Ενώ ο Μάρτιν Κάλαναν δεν είναι φιλόδοξος, έχει πολύ περιορισμένες φιλοδοξίες και συμμαχή με τους λιγότερο ικανούς. Δεν ξέρω ε, αν ε, θυμάστε ότι έχουμε βουλευτικές εκλογές στη Βρετανία σε ε, τρεις μέρες και το συντηρητικό κόμμα του Μάρτιν μιλάει για την πράσινη οικονομία, τα, ε, τις πράσινες θέσεις εργασίας και εμείς μιλάμε για το 2020 και τις θέσεις εργασίας της πράσινες μέχρι τότε. Στην πρόταση όμως που έχουμε ενώπιόν μας θα έλεγε ότι εδώ μάλλον την πάτησε, διότι αυτές είναι ανάδρομες προτάσεις. Είναι δηλαδή ένα χαστούκι στο πρόσωπο της βιομηχανίας. Αν γίνουν δεκτές, ε, συγγνώμη το λέω και προς το ΕΛΚ, δεν είναι φιλόδοξες προτάσεις και στο τέλος η Ευρώπη θα είναι λιγότερο αποδοτική. Στο τέλος οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα είναι πιο ακριβές από ό,τι πρέπει. Θα πληρώνουν περισσότερο για να κατασκευάζουν και να κυκλοφορούν τα οχήματα και αυτό θα συμβάλλει στη μείωση θέσεων εργασίας σε άλλες χώρες. Ε, ε, θα πρέπει να μην ακούσετε τα μεγάλα ονόματα των κατασκευαστών, αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να εξοικονομήσουν χρήματα από την κυκλοφορία των οχημάτων. Ε, μετά την Πέμπτη έλα, έλα ανανεωμένος, πιο φιλόδοξος και με καλύτερες προτάσεις. Σκέψτε το μετά. Κρίμα που είμαστε σε λάθος αίθουσα. Δεν υπάρχει web stream και δεν υπάρχει κανεί να μας ακούσει στα πέρατα τη γη τόσο ωραίε ομιλίε. Γιατί αυτά είναι προεκλογικές ομιλίε. Η επόμενη παρέμβαση. Ποιος είναι, ο Μπάς Άικοτα από τους Πράσινους. Εγώ. Ευχαριστώ. Πράγματι έχουμε εκλογές τον Ιούνιο. Έχουμε εκλογές τον Ιούνιο. Και οι Βέλγοι γενικότερα τους περιμένουν πολλές τέτοιες αναμετρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα ακολουθήσουν νέες εκλογικές ομιλίες. Άκουσα όμως προσεκτικά αυτά που είπε ο Κρίση γιατί πέραν του εκλογικού χαρακτήρα ε, το περιεχόμενό του ήταν πολύ σωστό. Τον ευχαριστώ λοιπόν. Για μας σαν πράσινος. βλέποντας την πρόταση αυτή, την οποία έκανε ο κύριος Κάνχαν, πράγματι νιώθουμε λίγο απογοητευμένοι. Πρόκειται για ένα déjà μια τέτοια αίσθηση Όποτε μιλάμε για αυτοκίνητα, για εμπορικά οχήματα, ξαφνικά ο πράσινος λόγος και η Ευρώπη του 2020 εξαφανίζεται γιατί έχουμε να κάνουμε με την κεντρική την βιομηχανία ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο κύριος Κάναχαν στην ουσία αυτό που κάνει είναι να καθιστά ασθενέστερους τους στόχους οι οποίοι είναι κρίσιμοι για να μετατρέψουν την οικονομία μας και να την κάνουν πιο οικοαποτελεσματική. Πράγματι συμφωνώ μαζί του ότι η βιομηχανία των Vans είναι πιο ε, χαρακτηριστική, είναι διαφορετική μάλλον από την ε, βιομηχανία που παράγει ιδιωτικά αυτοκίνητα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν διαφορετικούς στόχους. Και όταν μιλάμε για κυρώσεις και για το λεγόμενο pooling, τον συνδυασμό ή συνδυαστική χρήση, τότε ε, θα πρέπει να μην υπάρχει διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση τους. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει κάτι το ασύμβατο στις προτάσεις του εισηγητή. Διαφωνούμε λοιπόν με τις δηλώσεις του εισηγητή, σύμφωνα με τις οποίες ε, ότι θα πρέπει να υπάρχουν ε, ίδιες κυρώσεις αλλά διαφορετικοί στόχοι. Αν δει κανείς τη λογική της Επιτροπής για το πώς φτάνει στα επίπεδα των κυρώσεων, των προστήμων, το κάνει αυτό γιατί θεωρεί ότι είναι το ύψος που απαιτείται έτσι ώστε να περάσει σε πιο καινοτόμες μορφές παραγωγής. Δεν είναι τυχαία τα ποσά αυτά. Τα σκέφτηκαν τα ποσά αυτά γιατί πιστεύουν ότι λειτουργούν σαν κίνητρα για την καινοτομία. <coughs> Συμφωνούμε με τον εισηγητή ότι θα πρέπει να υπάρξει διαφορά στην αντιμετώπιση αυτοκινήτων και βαν. Και όπως είπε ο Chris Davis, αν δει κανείς τις μελέτες και δει την πληροφορία που κυκλοφορεί, το 2020 μπορεί σίγουρα να είναι ε, και πιο αποτελεσματικός από το 175 ή από το 135. Γι' αυτό είναι ανόητο να πούμε ότι πρέπει να μειώσουμε αυτή την αλλαγή των 50 γραμμαρίων σε, μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο γιατί θα μπορούσαμε να προτείνουμε να φτάσουμε τα 125. Λοιπόν, ελπίζω αυτά που λέει ο Καλχάν να υπακούν σε μια εκλογική, θα έλεγα, λογική και μια εκλογική τάση. Ελπίζω μετά τις 6 Μαΐου να διορθωθούν. Τώρα για τους κόφτες εδώ θα συμφωνήσουμε μαζί σας Συμφωνώ και με τον Ματίας ότι πράγματι είναι τεχνικά εφικτό και δεν θα πρέπει να ζητήσουμε 120 για τέτοια είδες οχήματα, θα πρέπει να φτάσουμε τα 100 χιλιόμετρα. Αυτό είναι από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους μείωσης της εκπομπής καυσαερίων και γι' αυτό το ΕΛΚ όταν κάνουμε τις προτάσεις μας και τις υποστηρίξεις θα δείξει ότι είναι και αυτό πράσινο. Ευχαριστώ. Η Ζαμπίνη θα μα πει περισσότερα ακόμα. Όχι, όχι, δεν θα βγάλω προεκλογικό λόγο. Διαφωνώ με τον κύριο Κάλαναν για τις οριακές τιμές. Είπε ότι είναι διαφορετικά τα επιβατικά, αλλά τα ελαφρά επαγγελματικά προσανατολίζονται λίγο και προς τα επιβατικά και τη δικιά τους τεχνολογία. Συχνά απλώ είναι διαφορετική η δομή τους, αλλά οι κινητήρε των επιβατικών πολλές φορές ε, ακολουθούν. Και οι εκπομπέ είναι τώρα 200 περίπου, ένα χιλιόμετρο, ε, γραμμάρια, ε, CO2. Νομίζω ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να, θέσει σαφή, να δώσει σαφή μηνύματα, μπορεί τεχνολογικά να έχουμε πρόοδο και τα 135 γραμμάρια που προτείνει η Κομισιόν μέχρι το 2020 δεν είναι καν αυστηρό στόχος για τους κατασκευαστές, δηλαδή είναι εφικτότατος. Και στο, και στο 125 μπορούν να πάνε το 2020. Είχε γίνει συζήτηση και των περιβαλλοντικών ενώσεων και ε, έλαβε χώρα κάποιος ένας, ε, έλαβε χώρα διάλογος και είπαν ότι βέβαια θα είναι λίγο πιο ακριβή η ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής και βέβαια αυτό θα μπει μέσα στην τιμή του αυτοκινήτου. Ο αγοραστής θα τα πληρώσει όλα αυτά. Αλλά γίνεται να μειώνονται οι εκπομπές. Επίσης ε, είπαμε 175 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο αυτό γίνεται και με την υφιστάμενη τεχνολογία. Η Volkswagen, η Renault, η Ford έχουν μοντέλα που καλύπτουν αυτές τις προδιαγραφές. Θα γίνει μια προσαρμογή στο μοντέλο και γι' αυτό το 2010 τέθηκε ο στόχος αυτός των 175 γραμμαρίων. Άλλη αναβολή δεν συζητείται καθόλου. Επίσης, Για τα επιβατικά ή χρειάζονταν φιλόδοξη νομοθεσία γιατί οι κατασκευαστές δεν ήταν διατεθειμένοι να κατέβουν στις εκπομπές ε, η δήλωση αυτοδέσμευσης δεν έδωσε καλά αποτελέσματα. Επίσης ο στόχος στα ελαφρά επαγγελματικά των 175 γραμμαρίων ήταν που γνωστός εδώ και καιρό δεν μπορούμε να, το, να έχουμε ε, άλλη αναβολή. Από το 2012 πήγαμε στο 2016, πρέπει να ε, επιτευχθεί ο στόχος και το δέχτηκε και η βιομηχανία. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία τώρα ε, εργάζονται βέβαια για να ανοίξουν παραθυράκια στην ομοθεσία δεν θέλω να εισαχθούν και, ή μάλιστα να αυξηθούν ή να χορηγούνται για μακρότερο χρονικό διάστημα αυτά τα super credits. Δεν έχει νόημα οχήματα που έχουν λιγότερο από 500 γραμμάρια να Ε, παραμείνουν ε, ε, περιορισμένα μονοχήματα θα πρέπει να επηρεαστεί όλος ο στόλος. Και εγώ είμαι υπέρ των κοφτών και στα 100 χιλιόμετρα όπως για τα φορτηγά. Αυτοί οι κόφτες είναι καλό πράγμα. Η Ford έχει αυτή την τεχνολογία για να τηρούνται και οι οριακές τιμές και αυτό οπωσδήποτε θα μειώσει τις εκπομπές. Όμως ε, δεν θα πρέπει να είναι εναλλακτική αντί, ε, η, λύση των κοφτών αντί για ε, αυστηρότερα, αυστηρότερες προδιαγραφές γιατί και αυτό το έχω ακούσει. Επίσης ε, είναι πολύ σημαντικό ο κανονισμός του 2013 να μην ε, ακολουθήσει ε, την πρόταση στην Κομισιόν σε σχέση με την ε, αξιολόγηση αντιχτή που των επιπτώσεων ε, και αυτό πάλι να οδηγήσει με τη σειρά του σε μια αποδυνάμωση των στόχων. Άπαξ δεν πρέπει μετά να αποδυναμωθούν. Ο Καρλ ο Φλόρενς. Ο Καρλ για τα αυτοκίνητα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ας αρχίσω με την ε, αυτοδέσμευση του 1997 που υποτίθεται ότι θα ίσχυε το 2007. Ήταν η μεγαλύτερη πολιτική ε, απογοήτευση ή κοροϊδία της πολιτικής μου ζωής. Και η τελευταία συζήτηση για τα αυτοκίνητα το είπε και ο πρόεδρος μόλις. Κοιτάξτε να δείτε. Διαβάστε λίγο την ανακοίνωση τύπου ε, της αυτοκινητοβιομηχανίας όταν άρχισε αυτό το θέμα να συζητείται. Ότι είχε χαλάσει ο κόσμος. Και κοιτάξτε τι λέγανε μετά το τέλος της συζήτησης και κοιτάξτε τι αυτοκίνητα αγοράζουμε σήμερα και κυκλοφορούν στην αγορά. Σας λέω ότι ακούω διάφορες ομιλίες εδώ σήμερα και το λέω πολύ συνειδητά. Φαντάζομαι ότι είναι παραμονές Χριστουγέννων όταν ήμουν μικρός. Γιατί και τότε είχαμε την ώρα του παραμυθιού αυτή. Κυρίες και κύριοι, η αυτοκινητοβιομηχανία για τους στόχους που τη ζητάμε από το 2012 μέχρι το 2015 έχει πετύχει ήδη σήμερα τους στόχους αυτούς σε ορισμένους τομείς. Οπότε δεν θα είχα εγώ αυτούς τους φόβους και τις αγωνίες ή να έλεγα ότι ε, όλοι οι κινητήρες που μπαίνουν σε ένα φορτηγάκι, Volkswagen, δεν ξέρω τι, ε, θα πρέπει να είναι ε, κινητήρες των ε, ε, φορτηγών. Όχι, ένα κινητήρα γκολφ κανονικό είναι ενό αλλού τύπου τη Volkswagen. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά αυτά που λέει ω αριθμητικά στοιχεία Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι καλά. Αν ε, μου ζητούσατε να αλλάξω εγώ ένα ε, αριθμητικό στοιχείο και μια οριακή τιμή, θα την έκανα πιο αυστηρή. Γιατί μόνο όταν του δίνει στόχου, τότε θα του πετυχαίνουν. Και αυτό μπορεί να σα εκπλήσει. Και σήμερα είναι. Και η απόδειξη. Μπορείτε να τη δείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα που πουλάει αυτοκίνητα. Γι' αυτό του στηρούν του στόχου, γιατί είναι δεσμευτικοί. Καλά, εγώ δεν θα υποβάλω αυστηρότερη τροπολογία, αλλά αν υπάρξει άλλη πλειοψηφία θα την υπερψηφίσω κι εγώ. Και εγώ, κυρίε και κύριοι, πρέπει να σα πω ότι μόνο εκείνο που. Ε, αγοράζει ε, τα πιο καθαρά αυτοκίνητα, μπορεί να τα πουλάει κιόλα. Μπορεί αυτό να είναι επώδυνο, να είναι δυσάριστο, αλλά θα πρέπει να το τηρούμε. Και κάτι άλλο, συμφωνώ με πολλού συναδέλφου έχει προβλήματα και αυτοκινητομηχανία και εγώ δεν το αμφισβητώ. Και ένα από τα προβλήματα είναι ότι η βιομηχανία πετρελαιοειδών ε, σήμερα έχει τέτοια εξουσία στον κόσμο που όσο καινοτόμο και να είσαι, σε παρεμποδίζει. Τα τελευταία 30 χρόνια είχε τη λιγότερη καινοτομία. Τα καύσιμα ήταν και παραμένουν ανιαρά. Δεν έχουν την παραμικρή καινοτομία. Είναι βαρετά τα καύσιμα, τα ορυκτέλα και τα πετρελαιοειδή. Και άμα του βάζει τέτοιο κάψιμο του κινητήρα, ε, ε, δεν είναι απορία άξιο που δεν είναι πιο ε, αποδοτικό δεν εξοικονομεί ενέργεια. Να πιέζεται και η ε, πετρελαιοβιομηχανία που δεν μπορούμε να την αναγκάσουμε και το ξέρω. Αλλά κοιτάξτε και πάλι τι λέγανε πριν την έναρξη τη συζήτηση για τα γεωταχή οι εταιρείε και κοιτάξτε τι λένε στο τέλο τη συζήτηση. Και δεν χρειάζεται να έρθει στη δική μου πολιτική ομάδα να πάμε στον Chris Davis, τα ξέρει και αυτός. Τι λέγανε και μετά τα ανερούσαν. Αν τα διαβάσετε αυτά θα καταλάβετε ότι δεν είμαστε σε κακό δρόμο. Συχνά, αρκετά συχνά επικρίνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τώρα δεν την επικρίνω ή λίγο μόνο. Ναι, έγινε πολύ μεγάλη φασαρία. Είναι τελείως διαφορετικό το πρόβλημα, αλλά γενικά έχουμε πολύ καλή συνεργασία και θα τα βρούμε. Ε, στο μέλλον ε, εύχομαι να έχουμε πολύ περισσότερο θάρρος. Ευχαριστώ. Ναι, η απογοήτευση ε, κρατάει χρόνια, μια ζωή ολόκληρη με την θελούσια δέσμευση και δεν πρόκειται να την ξεφορτωθείτε. Ήταν μια ενήλικη τοποθέτηση αυτή. Ο Βιτόριο Πρόντι, επόμενος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή μας, τον κύριο Κάλαναν, για την εργασία του. Όμως ε, έχω κάποια δυσκολία εδώ. Πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε ότι υπάρχουν ειδικοί κύκλοι δοκιμών αυτών των κατηγοριών ε, οχημάτων λόγω των ειδικών εργασιών που εκτελούνται με αυτά. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε πιο περιοριστικοί για τις εκπομπές. Ιδιαίτερα εις ό,τι αφορά τα όρια ταχύτητος. Θα μπορούσαμε να είναι αντιστρόφως ανάλογα προς το βάρος που μεταφέρουν τα οχήματα γιατί όσο υψηλότερη η γενικότερη μάζα τόσο μεγαλύτερη η ενέργεια που διαχέεται και που χάνεται στην επιτάχυνση και στην ε, πέδηση του συμβατικού οχήματος. Οπότε, ναι, τα όρια ταχύτητας πρέπει να είναι χαμηλότερα για τα βαρύτερα οχήματα. Υπάρχει νομίζω και ένα άλλο πρόβλημα. στην προσπάθεια ενθάρρυνσης του κόσμου να χρησιμοποιεί άλλων τύπων οχημάτων διαφοροποιώντας τα συμβατικά οχήματα. Μικρότερα ας πούμε οχήματα για μικρής κλίμακας δημόσιες μεταφορές ή συλλογή. Αν το δούμε αυτό, στις αστικές περιοχές διαπιστώνουμε ότι ήδη υφίσταται τεχνολογία για να εφοδιαστούμε με υβριδικά οχήματα και οι συνεχείς ε, επιταχύνσεις και παιδίσεις που υποχρεούνται να κάνουν τα οχήματα αυτά θα ήταν ιδεώδης όταν το αυτοκίνητο είναι υβριδικό και θα μειώνονταν οι εκπομπές γενικότερα και όχι μόνο το διοξίδιο και το διοξίδιο του αζότου και το μονοξίδιο του άνθρακα όλα θα μειωνόντουσαν οπότε αυτό είναι ένα πρόβλημα πρέπει να επιδείξουμε την τόλμη να προχωρήσουμε σε κίνητρα να πάμε σε υβριδικά τελείωση ή ηλεκτρικά οχήματα 100% πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, συμβουλεύσουμε τις, τους ΟΤΑ, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, να θέσουν όρια ταχυτήτων σε αστικές περιοχές που θα διασφαλίζουν μείωση και των αερίων του θερμο, θερμοκηπίου και τους οργανικούς ρηπαντές. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τις ε, τοπικές αρχές να περιορίσουν τον αριθμό των οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής κάψης στις αστικές περιοχές. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Η κυρία ε, um, Ευχαριστώ. Σαφές είναι ότι οι οδηγίες, οι φιλόδοξες ε, ε, οδηγίες για το περιβάλλον είναι καλές και για την καινοτομία και για την απασχόληση. Δεν είναι απειλή. Είναι ευκαιρία οι φιλόδοξες οδηγίες και αποδείχθηκε αυτό από τον κανονισμό για τα αυτοκίνητα. Γιατί έδειξε ο υπολογισμός ότι η αυξημένη απόδοση καυσίμων επετεύχθη πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν. Και το είπαν αυτό οι προηγούμενοι ομιλητές. Πιστεύω λοιπόν γι' αυτό ότι θα πρέπει να πιέσουμε για πιο φιλόδοξους στόχους. Από 175 το 2016 μπορούμε να περάσουμε στο 160. Να, να κατέβουμε από το 175 στο 160 για το 2016. Η εναρμόνιση λοιπόν μεταξύ, χρονικά, με, μεταξύ αυτού του ε, νομοθετήματος και του άλλου για τα αυτοκίνητα θα ήταν καλό. Το ίδιο ισχύει και για το 2020. 125 γραμμάρια είναι εφικτός στόχος και αυτό είναι 38% μείωση σε σύγκριση με τα παρόντα επίπεδα και αυτό θα ευθυγραμμιζόταν καλύτερα και με το στόχο για τα αυτοκίνητα που είναι 40% η μείωση εκεί για τα αυτοκίνητα μέχρι το 2020. Τώρα, για τα όρια ταχύτητα και τους κόφτες, ε, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ φιλόδοξοι στα όρια ταχύτητας στον περιορισμό της ταχύτητας και νομίζω ότι θα πρέπει να ταχθούμε, εγώ τάσομαι τουλάχιστον υπέρ του φιλοδοξότερου στόχου. Ευχαριστώ. Η κυρία Λαπάζ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κάλαναν για την έκθεσή του. Οι προτάσεις του ε, ακριβώς αυτό θέλουν να περιορίσουν ε, την εκπομπή των καυσαερίων. Ξέρω ότι έχει γίνει μεγάλο λόμπινγκ και για τα χρονικά όρια και για τις οριακές τιμές και τις προδιαγραφές. Είναι μια στρατηγική ε, που είναι γνωστή και έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως και τελικά είναι αρκετά αντιπαραγωγική. Αν δούμε σήμερα τι προτάσεις κάνει η κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία. Έχουν μικρά οχήματα, ηλεκτροκίνητα. Και τι προτείνει η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Θα λέγαμε ότι καλά θα κάναμε πριν από λίγα χρόνια να είμαστε πολύ πιο απαιτητικοί και θα ήμασταν τότε εμείς ηγέτε σε αυτά και όχι το κινέζικο αυτοκίνητο. Ε, δηλαδή, θα πρέπει να δίνουμε κίνητρα, να βάζουμε τέτοια πρότυπα και προδιαγραφέ που να είναι μια όθηση. Ε, και το είπαν και άλλοι συνάδελφοι, οι τεχνολογίες υπάρχουν, Αλλιώ είναι αντιπαραγωγικό και για το περιβάλλον αλλά και για τη βιομηχανία και τις θέσει απασχόληση. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Συμφωνώ απολύτω με αυτά που προτείνουν οι συνάδελφοι. 160 γραμμάρια για 2014-2016 και 120 όχι 135 για το 2020. Σε ό,τι αφορά τώρα τα πρόστιμα για το 2014 με 2018 ας προσπαθήσουμε να απλουστεύσουμε λίγο το σύστημα και να αναθεωρήσουμε δεχομένως κυρώσεις και τα πρόστιμα για τα ε, οχήματα που ε, εκπέμπουν ε, πολλά καυσαέρια, πολύ διοξείδιο του άνθρακα, πάνω από 15% της ανώτατης ε, τιμής. Και επίσης θα πρέπει να πηγαίνουν και στην κατηγορία N2 και M2, που είναι μίνι μπας και μη φορτηγάκια, και ακριβώς πάντα στα πλαίσια της διαφάνειας και της ενημέρωσης που θέλουμε να διαφημίζονται τα αυτοκίνητα που καλύπτονται από τη βιομηχανία. Δηλαδή να λέμε ποιες είναι οι ενεργειακές επιδόσεις και οι εκπομπές ε, των διαφόρων οχημάτων. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ, Ρίχαρτ Τσέπερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Στην τελευταία συζήτηση ε, είπα στην Κομισιόν ότι σε αυτό το τομέα θα μπορούσαμε να δούμε τις διαφορές ε, και να τις επεξεργαστούμε καλύτερα μεταξύ επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών. Πάντως η πρόταση είναι καλή και δεν έχει σημασία τώρα το 175, 180, 160. Το σημαντικό είναι ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, προγραμματισμός ενός σημαντικού τομέα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Δεν θα μιλήσω πολύ υπέρ της μιας ή της άλλης κατεύθυνσης, αλλά χρειάζεται ένα πλαίσιο πέρα από τις εκλογές γιατί η αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη έχει μεγάλη δυνατότητα να είναι μακροπρόθεσμη επιτυχής και ανταγωνιστική. Δίνει και πολλές θέσεις εργασίας. Να υπάρχει ένα πλαίσιο λοιπόν το οποίο θα ανταποκρίνεται σε, πιθανές, ε, σε πιθανή ανάπτυξη ώστε να φτάσουμε κάποια στιγμή σε μία ε, εποχή που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους μειούμενους σπόρους. Ε, είναι σημαντικό να προβλέψουμε. Αυτά τα οχήματα θα πρέπει να συνεχίσουν να αγοράζονται, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά σε όλο τον κόσμο, όπως και στο παρελθόν. Άρα λοιπόν εκεί εστιάζομαι, στον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό. Πολύ συνειδητά λέω ότι δεν πρέπει να ε, περιοριστούμε μόνο σε εκπομπές του σιωτού. Υπάρχουν και άλλες εκπομπές. Αν έχουμε υποχρεώσεις μόνο σε αυτό το θέμα, μπορεί να αυξηθούν τα διοξίδια του θείου, του αζότου και αυτό δεν είναι καλό για το περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Οπότε νομίζω ότι αυτά τα θέματα που έβαλε και η κυρία Βάις ε, Γκέρμπερ για τα super credit, για τις ε, ε, οικοκαινοτομίες να τις δούμε γιατί έτσι θα βελτιώσουν τη θέση μας γιατί αν επικεντρωνόμαστε έτσι ξεροκέφαλα στα γραμμάρια μόνο του διοξιδίου του άνθρακα δεν κάνει δεν είναι σωστό αυτό. Ε, το τυπικό 170 ή 175 δεν είναι τόσο σημαντικό. Σημαντικό είναι να δούμε πώς θα κινείται στους δρόμους ε, το αυτοκίνητο αυτό. Γι' αυτό η συζήτηση και σε άλλα φόρα. Δεν είναι τόσο σημαντική για να πέσουμε πάνω στον αριθμό και να επιμένουμε εκεί, αλλά να δούμε μακροπρόθεσμα πού κινούνται τα πράγματα. Ευχαριστώ. Η Κρίστα Κλάς. Ευχαριστώ πολύ. Παρακολουθώντας τη συζήτηση, ε, είδα ας πούμε σαν να έχουμε εδώ πέρα στο πόκερ να στοιχηματίζουμε και να βάζουμε τους πόντους μας ο ένας παραπάνω, όλος παρακάτω. Πρέπει να έχουμε ρεαλιστικούς στόχους, αυτό είναι το σημαντικό. Δεν έχει νόημα δηλαδή να πετάμε αριθμούς ε, ή να τους γράφουμε. Μιλάμε για μικρά επαγγελματικά οχήματα, και γι' αυτό τρομάζω λίγο ακούγοντα για κόφτες και περιορισμούς ταχύτητας και όρια. Ποιος τα οδηγεί αυτά τα αυτοκίνητα. Αν το δούμε και αυτό, βλέπουμε ότι είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι βιοτεχνίες που θα, ή τη μικρή που θα βάλουν το ζώο το, ή, θα βάλουν τους βοηθούς. Ε, αυτή η μικροί ας που θα πάνε για το κρασί θα, ε, ε, είναι κακό, θα είναι πολύ ώρα στο δρόμο αν δεν μπορούν να τρέξουν παραπάνω και αυτό βεβαίως ε, έχει αντίχτυπο και στο, στο χρόνο οδήγηση και στα εισδαπάνες ο συνάδελφος πρώτη είπε ότι κάποιος που ένα αυτοκίνητο, ένα τέτοιο επαγγελματικό το οποίο ε, μεταφέρει μεγάλα βάρη, έχει διαφορετική ε, κατανάλωση ενέργειας όταν επιταχύνει, όταν ε, φρενάρει. Επίσης ο χρόνος οδήγησης είναι πολύ σημαντικός αυτά, θα πρέπει να τα δούμε για να σταθμίσουμε κόστος ωφέλεια και να... Είναι ένα επιχειρήμα απλώς, ένα επιχείρημα και η μείωση της, της ταχύτητας. Ε, σίγουρα δεν πρέπει να περιοριζόμαστε σε αριθμούς μόνο να μειώσουμε την ταχύτητα δεν ε, κάνουμε τίποτα. Ε, οι δαπάνες και η επιβάρυνση εκφράζονται μέσα από αυξημένους χρόνους οδήγησης. Οπότε μην περιοριζόμαστε σε έναν αριθμό, αλλά θα πρέπει να δούμε με ευρύτερο πνεύμα, πιο ανοιχτό ορίζοντα όλο το ζήτημα. Όπως είπε και η κυρία Βάις Γκέρμπερ. Ε, με τις γραπτές της και με την παρέμβασή της εδώ. Πρέπει δηλαδή να έχουμε ένα ευρύτερο πνεύμα στην προσέγγισή μας. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή ήταν η τελευταία παρέμβαση αναμφίβολα πρέπει να είναι πιο καθαρός ο τομέας των μεταφορών και εις ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και τη μεγαλύτερη συμβολή του στην προστασία του κλίματος. Δηλαδή οι εκπομπές του CO2 πρέπει δραστικά να μειωθούν όπως προφανώς και οι άλλοι ρήποι, διοξίδια του θείου, του αζότου, ιδιαίτερα στους, ε, στον αστικό χώρο. Βεβαίως υπάρχουν κάποιοι αριθμοί που πέφτουν πάνω στη ζυγαριά 125, 130, 175, 150 ε, θα τα ξαναδείτε ο καθένας από σας ε, για να δούμε τι επιπτώσεις έχουν όλα αυτά. Ο Μάρτιν Κάλαναν ε, άκουσε πολλά σχόλια, το λέω διπλωματικά, από πολλές πλευρές. Σίγουρα υπάρχει μια ε, διαφορά μεταξύ επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών γιατί τα επιβατικά είναι 50% δίζελ ενώ το, τα επαγγελματικά ελαφρά είναι 90% δίζελ ε, το καύσιμο. Οπότε ε, με το πέρασμα έχουμε διαφορά. Περνάμε στο δίζελ από τη βενζίνη και το δίζελ είναι καλύτερο και ε, υπήρξαν και πολύ μεγάλες πρόοδοι ό,τι αφορά τη διαδικασία της κάψης. Αυτά τα άλματα δεν τα περιμένουμε πια, τελείωσαν στον τομέα των ελαφρών επαγγελματικών, αφού το 90% ήδη πέρασαν στον διζελ. Αυτά μεταφέρουν βάρη. Και υπάρχουν διάφορα μεγέθη. Ο ένας βιοτέχνης έχει μικρότερο γιατί έχει μικρότερες ανάγκες μεταφοράς, ο άλλος έχει μεγαλύτερο κουβαλάει περισσότερα. Ε, Επίση ρημουλκούν και βάρη, φορτία ε, και στο τεχνολογικό άλμα που ανέφερε και ο Ματίας θα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν ε, δυνατότητες να υπερβούμε κάποια όρια. Δηλαδή ε, μπορεί να περάσουμε μετά σε μπαταρία ή σε υδρογόνο ή σε υβριδικό και θα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν μπαταρίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλα οχήματα πέρα από τα επιβατικά. Γιατί τώρα έχουμε κάτι πολύ μεγάλα οχήματα τα οποία ε, ε μεταφέρουν 150 τρέχουν 150-200 χιλιόμετρα. Α, ε, ή τα επιβατικά που φτάνουν μέχρι 300 χιλιόμετρα. Αλλά ε, επίση παίζει ρόλο και η, ε, ε διάρκεια ζωής, ο, ο κύκλος ζωής του ε, οχήματος, ε, αν μεταφέρουν φορτία και την επιχείρηση. Ε, αυτό οπωσδήποτε επηρεάζει και τη διάρκεια ζωή του οχήματο. Ο εισηγητή τώρα έχει το λόγο. Ο Μάρτιν Κάλαναν. Α, όχι. Πριν δώσω η Κομισιόν. Η Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον κύριο Κάλαναν για το σχέδιο έκθεσης. Ευχαριστώ και τους σκιώδεις εισηγητές. Θα ήθελα καταρχήν να μιλήσω για μια ευρύτερη εικόνα, γιατί όπως είπατε είναι μεγάλος τομέας αυτός των μεταφορών, ο οποίος ευθύνεται για μεγάλο ποσοστό αερίων θερμοκηπίου και αν ε, πετύχουμε το στόχο μέχρι το 2020 και μετά μέχρι το 2050, σημαντικό είναι να έχουμε φιλόδοξες πολιτικές και νομοθεσίες από πριν ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε τους φιλόδοξους στόχους. Αυτή η πρόταση για τα ελαφρά επαγγελματικά είναι μέρος της πρότασης και οπωσδήποτε μελετήσαμε προσεκτικά και τα στοιχεία, τα αριθμητικά, τα νούμερα και υπάρχουν και μελέτες επιπτώσεων που τα στηρίζουν. Γι' αυτό σε αυτό το στάδιο η Κομισιόν πιστεύει ότι οι στόχοι του 100, των 175 το 2016 και το 135 το 2020 είναι εφικτοί στόχοι και ρεαλιστικοί. Γι' αυτό λοιπόν ε, είμαι γνώμων για τα 175, στον κύριο Κάλαναν δηλαδή που τα θέλει. Πιστεύω ότι και μακροπρόθεσμα θα πρέπει να είμαστε ανάλογα ε, φιλόδοξοι τα 125 έδειξε μια μελέτη επιπτώσεων, τα 125 γραμμάρια, ότι είναι εφικτός με τις ε, βελτιώσεις στην τεχνολογία και το εξετάσαμε αυτό, όμως ε, καταλήξαμε στα 135 για το 2020 που είναι ε, φυκτός και φιλόδοξος ταυτόχρονα στόχος και νομίζω ότι αυτό είναι ο στόχος ε, στον οποίο εμένει ναι, η Κομισιόν τώρα. Διάφορα θέματα έθεσαν τα μέλη της Επιτροπής σας, για παράδειγμα τις κυρώσεις. Γιατί ένα πρόστιμο να είναι υψηλότερο για τα επαγγελματικά από ότι για τα επιβατικά. Το εξετάσαμε πολύ προσεκτικά και η ανάλυση επιπτώσεων έδειξε ότι ο οριακό κόστος συμμόρφωση για τα Βάν είναι 130 ευρώ και όχι 95 ευρώ αναγραμμάριο όπως τα αυτοκίνητα. Οπότε υπάρχει ένα οικονομικό σκεπτικό, υπάρχει μια λογική. Δεν είναι δηλαδή ότι ένα γραμμάριο σιωτού είναι πιο ακριβό για τα βαν, αλλά το οριακό κόστος συμμόρφωσης παίζει ρόλο. Είναι πιο καλό να ε, οι κατασκευαστές να συμμορφωθούν έτσι προς την νομοθεσία από ότι όχι. Επίσης, τα super credits. Για παρόμοιο λόγο εφαρμόθηκαν γιατί έτσι ε, προχωρεί η καινοτομία. Αυτό ε, μας αφορά πολύ στην νομοθεσία και στη στρατηγική της Ευρώπη για το 2020 είναι σημαντικό να γίνει σε όλη τη βιομηχανία καινοτομία, πολλές καινοτομίες και στην αυτοκινητοβιομηχανία, ούτως ώστε να παραμείνει ο τομέας αυτός ανταγωνιστικός ε, με ε, ε, σε σχέση με τους άλλους εταίρους μας εκτός Ευρώπης. Φιλόδοξη αλλά και προσεκτική στη χρήση τους των super credits, γιατί αν έχουμε ένα Ε, γιατί ανάλογα με τον κινητήρα ή και την, ε, την ε, εκπομπή θα χρησιμοποιούνται. Χρειάζονται να εφαρμόζονται με προσοχή τα super credit, αλλά αναγνωρίζουμε το καινοτόμο δυναμικό τους. Τώρα, για τους κόφτες, ε, αναφέρεται και στις αιτιολογικές σκέψεις της πρόταση της Κομισιόν. Χαίρομαι που βλέπω τον ενθουσιασμό για τους κόφτες στην Επιτροπή αυτή και στην Επιτροπή Μεταφορών επίσης γιατί υπάρχουν αποδείξεις. Ξέρω ότι το, οι Επιτροπές Περιβάλλοντος ε, και Μεταφορών έχουν ασχοληθεί με το θέμα και φαίνεται ότι οι κόφτες μειώνουν τις εκπομπές των φορτηγών και έχουν και άλλα δυνητικά ωφέλη όπως βελτιώνουν την οδική ασφάλεια κλπ. Τώρα για το πούλινγκ. Ε, εξέτασα προσεκτικά την πρόταση του εισηγητή για το πούλινγκ και οπωσδήποτε βλέπω τα πλεονεκτήματα για εκείνους τους ε, κατασκευαστές που ε, κατασκευάζουν και ελαφρά φορτηγά και επιβατικά. Οπωσδήποτε ε, είναι σε μειονεκτική θέση οι κατασκευαστές που φτιάχνουν μόνο μια κατηγορία από οχημάτων και όχι την άλλη. Θα συζητήσω με τον εισηγητή για να δούμε την πρακτική εφαρμογή αυτής της ιδέας, γιατί θα πρέπει να το σκεφτώ λίγο παραπάνω πριν καταλήξω σε μια εμπεριστατωμένη γνώμη. Καταρχήν όμως η έννοια του pooling μεταξύ επιβατικών ε, επαγγελματικών λαφρών δεν είναι ξένη ιδέα. Σίγουρα το λαμβάνουμε υπόψη μας ε, στα πλαίσια της πρότασης, αλλά να δούμε τις πρακτικές επιπτώσεις. Είναι μια ιδέα η οποία είναι θετική και πρέπει να εξεταστεί περισσότερο. Τέλος, διάφορα μέλη μίλησαν για τα λεγόμενα πολυφασικά αυτοκίνητα multi-stage. Η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι είναι δύσκολο ο τομέα και γι' αυτό έχει ε, συντάξει non-paper για τη γραμματεία και του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και εκεί αναφέρεται μία πρόταση στο σχέδιο έκθεσης από την Επιτροπή Μεταφορών. Ε, σε σχέση με τα πολυφασικά λοιπόν έχουμε τρόπο να ε, λύσουμε τα προβλήματα αυτά. Και τέλος θα ήθελα να πω ότι θα περιμένω με ενδιαφέρον τις ε, τροπολογίες σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής του. Και εγώ ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα σχόλιά της, λέει ο εισηγητής. Και όλα τα, μέρη, τα μέλη τα οποία πήραν λόγο μου έδωσαν χρήσιμες απόψεις. Κάποιες σύντομες απαντήσεις. Πρώτον, Σα σας ευχαριστώ για τη γενική σας υποστήριξη. Συμφωνώ με τα σχόλια που κάνατε και για τα κίνητρα. <clears throat> Το καρότο είναι καλύτερο από το μαστίγιο, συστηματικά. Και έτσι θα πρέπει να προωθήσουμε τα super credits και να δώσουμε θετικά κίνητρα στους κατασκευαστές για την παραγωγή πιο πράσινης τεχνολογίας. Γκρούτα, ευχαριστώ και εγώ για τα σχόλιά σας. Με μπερδεύετε με τον Λάγκεν. Εγώ δεν πρότεινα 140 μέχρι το 2025. Με έχουν συγκρίνει με πολλούς, αλλά όχι με τον Λάγκεν. Νομίζω ότι διαβάζετε πολλές ε, εκθέσεις και αυτό που είπατε για μένα δεν ανήκει σε μένα. Davis. Um, I have a, I, I probably hasn't realised it, but he's actually in Belgium at the moment. It's not an election on here. And most people in this room don't have votes, Chris, so I think... Οι εκλογικές ανησυχίες του κυρίου Ντέιβις ε, πηγαίνουν χαμένες, γιατί οι περισσότεροι εδώ δεν ψηφίζουν στις εκλογές η πρόταση την οποία κάνει είναι αυτή την οποία και εμείς ε, προτείνουμε μέχρι το 2020. Πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι ε, πάντως προσπαθώντας να το πετύχουμε αυτό, όχι σαν τους φιλελεύθερους οι οποίοι επιδιώκουν μόνο το βραχυπρόθεσμο εκλογικό κέντρο με τους ε, πράσινους. Είπε ότι είμαι εκλεκτός συνάδελφος και κατάλαβα ότι σαν εισαγωγή μετά θα ακολουθούσε η κατάπτωση για μένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει ε, εκτός από το θέμα του κόφτη ταχύτητα δεν συμφωνούμε στα διάφορε στις διάφορες τροπολογίες. <clears throat> Τελικά πολλοί από τους παραγωγούς βαν στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Η αγορά έχει πέσει, έχει πέσει κατά 30 με 40% τον τελευταίο χρόνο. Πάρα πολλοί απολύονται, υπάρχουν πολλές απολύσεις. Ελπίζω η αγορά να ανακάμψει λογικά, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε να μην επιβαρύνουμε τις επιχειρήσεις αυτές με υπερβολικές ρυθμίσεις. Νομίζω ότι πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι φιλόδοξη, ίσως υπερβολικά φιλόδοξη. Προτείνουν μία μείωση 10 γραμμαρίων κατέτος από το 2015 μέχρι το 2020. Λοιπόν, Κάποιοι άλλοι επιδιώκουν μεγαλύτερες φυσικά μειώσεις στον τομέα των εμπορικών οχημάτων, των ελαφρών εμπορικών οχημάτων. Αν και εκεί ξέρετε ότι υπάρχει θέμα μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων με μεγάλο βάρος και γι' αυτό οι προτάσεις τις οποίες κάνω εγώ παραμένουν με φιλόδοξες αλλά είναι και πιο ρεαλιστικές και θα οδηγήσουν τη βιομηχανία στη σωστή κατεύθυνση και θα υπάρξουν πολλές τροπολογίες από πλευρά των μελών και στο τέλος θα καταλήξουμε σε μια λειτουργική πρόταση και ευχαριστώ όλο τον κόσμο για τα σχόλιά του. Ευχαριστώ πολύ Μάρτιν Κάλλον για τα σχόλια αυτά. Για να ξεφύγουμε από τις Βρετανικές εκλογές βάλαμε την προθεσμία για τις τροπολογίες μετά την 6η Μαΐου. 10 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι λίγη. Οπότε μπορείτε όλοι να κάνετε τις ροπολογίες σας με την ησυχία σας και μετά τις 6 του μηνός με το καλό. Λοιπόν, ωραία. Some jokes are quite well in the debate that is... Δεν πειράζει να ελαφρύνουμε και λίγο τη συζήτηση, να λέμε και κανένα αστεάκι, μην είμαστε υπερβολικά σοβαροί. Επόμενο θέμα. Δίκαιο εισόδημα για τους αγρότες. Βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη. Κάνουμε εμεί γνωμοδότηση εδώ για την Επιτροπή Γεωργία. Η συγκήτρια είναι η κυρία Εστέρ Ραν Γκαρσία. Και τη δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όντω. Σχέδιο γνωμοδότησης καλούμαστε να εξετάσουμε που έχει εκπονηθεί για την καλύτερη λειτουργία της αλυσίδα, τροφικής Αλυσίδα. Τα ξέρετε κυρίως εσείς που έχετε μεγαλύτερη σχέση με τη γεωργία ότι εδώ και καιρό οι καταναλωτές, οι παραγωγοί κυρίως του πρωτογενού τομέα και οι καταναλωτές, οι οργανώσεις τους κάνουν ε, προτάσεις και αιτήσει για βελτίωση της τροφικής αλυσίδας. Πέρσι, στα τέλη του έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίδια κατέθεσε μια μελέτη που δεχόταν τις καταγγελίες αυτές όσο σωστές και έλεγε ότι υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, το πρώτο που κάνει τώρα η Επιτροπή και η γνωμοδότησή μου είναι να διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει το υπάρχον πρόβλημα. Και το δεύτερο που θέλουμε να κάνουμε με τη γνωμοδότησή μας είναι να δώσουμε ασφάλεια και ε, ωφέλεια και ισορροπία στους παραγωγούς και στους καταναλωτές και στο σύνολο της αγοράς. Και κάνουμε διάφορες προτάσεις λοιπόν για διάφορα μέτρα. Τι θέλουμε, τι ζητούμε, άμεσο συσχετισμό της τιμής που καταβάλλεται στον παραγωγό και της τιμής του καταναλωτού όταν φτάνουν τα προϊόντα. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε να μειώνονται ε, τα εισοδήματα των ε, παραγωγών, αλλά αυτό δεν αντανακλάται και στην τιμή καταναλωτού. Επίσης, προτείνουμε να έχει ε, η Ευρώπη κοινή στρατηγική για να βελτιώνει τη διαπραγματευτική δυνατότητα κάποιων κρίκων της αλυσίδας που είναι πιο αδύναμοι από άλλους. Αυτοί οι κρίκοι τι χρειάζονται. Να αλλάξει η ευρωπαϊκή νομοθεσία λοιπόν σε θέματα ανταγωνισμού και να εναρμονιστούν οι δράσεις των εθνικών αρχών ανταγωνισμού και να υπάρχει ειδική μέρημνα για το γεωργικό τομέα. Γιατί η γεωργία έχει ιδιάζουσα λειτουργία, λειτουργεί διαφορετικά από τους άλλου κλάδου οικονομία και θα πρέπει να το ξέρουμε αυτό στον ανταγωνισμό. Επίσης ζητείται μια καταγραφή των καταχρηστικών ε, πρακτικών. Στην αγορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι υπάρχουν καταχρήσεις στην αγορά, όπως είναι ε, διάφορες ε, προμήθειες ε, στην πώληση ή πώληση με ζημίες και άλλες επιβλαβείς πρακτικές. Θα πρέπει αυτά ρητά να απαγορεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπάρχει μια δημόσια λίστα των υπηρεσιών και των επιχειρήσεων που παραβιάζουν την νομοθεσία. Επίσης, θα πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται με τα προβλήματα στις πληρωμές, τους κακοπληρωτές. Μεγάλες αλυσίδες διανομής ε, μήνες μέχρι και χρόνια κάνουν ε, να πληρώσουν τους προμηθευτές τους και ε, οδηγούνται σε πτώχευση ορισμένοι προμηθευτές μεγάλων αλυσίδων διανομής. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να ενισχυθεί στην νομοθεσία, υποχρεωθούν αυτές οι εταιρείε να συμμορφώνονται στις ε, ε, περιόδους αυτές και να μην υπερβαίνουν το 12 μήνο. Επίσης να βρούμε κάποια μέτρα για να αποφύγουμε αθέμητες πρακτικές στην ανταγωνιστικότητα. Γιατί ο, μεγάλος παραγωγός και ο μικρός παραγωγός δεν είναι στην ίδια μοίρα. Ε, ε, ε, μια μικρή εκμετάλλευση, μια μικρή εταιρεία, ένας μικρός παραγωγός, ένα μικρό μαγαζί δεν έχει τις ίδιες αντιστάσεις με τους μεγάλους. Έτσι είναι ο βιομηχανικός ιστός και θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Και, ε, και επίσης θεωρείται ε, απαραίτητη μεγαλύτερη ολοκλήρωση ακριβώς και ε, διασύνδεση σε επαγγελματικές ενώσεις, ε, οι διάφοροι κλάδοι παραγωγής, στάνταρ συμβάσεις, εθελοντικές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα ευπαθή προϊόντα, ε, τα κράτη-μέλη να ζητούν, να απαιτούν να ε, γίνονται σεβαστές ρυθμίσεις. Αυτά τα σημεία, έξι σημεία, γνωμοδότηση είναι στο κάτω-κάτω. Ελπίζω να μου κάνετε προτάσεις για να εμπλουτίσω και εγώ τη γνωμοδότηση αυτή. Ευχαριστώ. Ε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ράνς, Γκαρσία λέει Και τώρα το λόγο έχει ο Τσάμπα Ταμπάιτζη. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εξ ονόματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, στην γνωμοδότηση αυτή θεωρούμε πολύ σημαντικά αυτά που λέει η συγκήτρια, για διάφορους λόγους. Υπάρχουν τρεις στοιχές πάρα πολύ σημαντικές για μας που ε, είμαστε Επιτροπή Περιβάλλοντος, έτσι, που αφορούν την Επιτροπή Περιβάλλοντος ασφάλεια τροφίμων, προστασία περιβάλλοντος. Πώς θα μεταφραστούν στη νέα γεωργική πολιτική. Είναι πολύ σημαντικά αυτά για μας. Το εισόδημα των αγροτών, πώς θα είναι εξασφαλισμένο, πώς θα μπορούν οι αγρότες να επενδύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, γιατί είναι παράγον κλειδί το περιβάλλον και θα είναι και στη νέα γεωργική πολιτική από το 2014 και μετά κυρίως. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος λοιπόν ε, ε, ενδιαφέρεται άμεσα γιατί την αφορά αυτό το θέμα. Το δεύτερο. Η δημιουργία τροφίμων. Η παραγωγή μάλλον τροφίμων και η κατάλωση ενέργειας για την παραγωγή τροφίμων. Δεν θα πρέπει τα τρόφιμα να ταξιδεύουν χιλιόμετρα, αποστάσεις είμαστε πάρα πολύ σπάταλοι στην κατανάλωσή μας και πολλά καυσαέρια εκπέμπονται όταν κυκλοφορούν τρόφιμα ε, χιλιάδες ε, χιλιόμετρα και μεταφέρονται από το ένα μέρος της Ευρώπης σε ένα άλλο. Θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε πάρα πολλές εκπομπές καυσαερίων και αερίων του θερμοκηπίου. Πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό επίσης κάτι άλλο. Τι γεωργία θέλουμε. Εντατική ή εκτατική. Αυτό πρέπει να το λύσουμε. Χρησιμοποιούμε ε, πάρα πολλά ορυκτά καύσιμα και καταναλώνουμε πόρους ε, που εισάγουμε, που δεν παράγουμε στην Ευρώπη. Καταναλώνουμε πάρα πολλές πρώτες ύλες, τις οποίες επίσης φέρνουμε από πάρα πολύ μακριά. Γι' αυτό είμαι ακράδαντα πεπισμένος ότι η έκθεση Μποβέ, που είναι πολύ σημαντική, ε, χρειάζεται και τη δική μας παρέμβαση. Συμφωνώ πολύ με την κυρία Εράντς και πρέπει να σκεφτούμε ότι η ανταγωνιστικότητα και ο ανταγωνισμός δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τον παγκόσμιο ανταγωνισμό ή τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό. Συμφωνώ και με τον Επίτροπο Τσόρο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο τοπικός ανταγωνισμός, να πολλούνται τα προϊόντα κοντά στον τόπο παραγωγής, να υπάρχει ανταγωνιστικότητα και ε, εντόπια και χώρια και μπορούμε εμείς να συμβάλλουμε σε αυτό για να μειωθούν τελικά τα καυσαέρια, τα αέρια του θερμοκηπίου. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή της ηγήτριας στο εξή. Συμφωνώ εγώ με τον Ζωζέ Μποβέ ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξει τις ρυθμίσεις για την ασφάλεια των τροφίμων. Διότι δεν μπορούμε να έχουμε τις ίδιες απαιτήσει από ένα μικρό σφαγί, ας πούμε, ή από μια μικρή εκμετάλλευση, τις ίδιες και ε, όπως ε, σε μια μεγάλη εκμετάλλευση ή σε ένα μεγάλο σφαγείο. Είναι πολύ σημαντική η ασφάλεια τροφίμων στην Ευρώπη. Υπάρχουν πολλές μεγάλες εταιρείες που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσει και εμεί βάζουμε τις ίδιες απαιτήσει στους μεγάλους και στους μικρούς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να αναθεωρηθεί. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν σοσιαλιστές συμφωνούν να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα εποπτείας και παρακολούθησης ασφάλειας τροφίμων, να συσταθεί αυτή η υπηρεσία με ιστοσελίδα επίσης, έτσι ώστε να κάνουν αιτήσεις εκθέσεις η παραγωγή τροφίμων για την ασφάλεια τροφίμων και να κυκλοφορούν αυτά δημόσια. Έχουμε και αρχές ανταγωνισμού, δεν αρκεί όμως. Στην Ουγγαρία πρόσφατα είναι ένα νόμο που ορίζει αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο. Και είναι ο ίδιος οργανισμός που ε, διαχειρίζεται και τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Λοιπόν, αυτός ο οργανισμός που δίνει τα χρήματα ε, ελέγχει και την ποιότητα. Και κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να κάνει ε, καταγγελία μέχρι και μήνυση αν διαπιστώνει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Νομίζω ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί και ένας τέτοιος ευρωπαϊκός οργανισμός για την Ένωση, όχι για ε, το κάθε κράτος ξεχωριστά. Στην ευρωπαϊκή νομοθεσία υπάρχουν διάφοροι τομεί στου οποίου δεν είμαστε αρμόδιοι εμεί βέβαια, αλλά η βιομηχανία, η Επιτροπή Βιομηχανία. Εξ ονόματο τη ομάδα μου θα πω επίση ότι θέλω να κάνω τροπολογίε για το θέμα αυτό διότι όλα αυτά που συζητούμε έχουν πτυχές και περιβαλλοντικές και που μας αφορούν και μας. Αυτά. Καλή γνωμοδότηση και ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Merci. Euh, Marie Tack, fru ordförande. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκαρσία για, την κυρία Γαρσία για μια εξαιρετική γνωμοδότηση. Είδα και τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και νομίζω ότι δεν καλύπτουμε το σύνολο της τροφιμικής αλυσίδας. Ξεχνάμε σαν παράδειγμα τον τομέα των προμηθειών, έναν τομέα ο οποίος μερικές φορές είναι δραστηριός ακόμα και πριν φτάσει κανείς στη γεωργική παραγωγή και στη γεωργία γενικότερα. Οι γεωργοί αντιπροσωπεύουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία αν τη συγκρίνει κανείς με τις εταιρείες, τις επιχειρήσεις οι οποίες αναλαμβάνουν ε, ε, ό,τι άλλο έχει σχέση με την αλυσίδα της διατροφής και αναφέρομαι εδώ στις, στα σπορία, στα χημικά, στα συντηρητικά, στις μεταφορές των προϊόντων. Ε, είναι πολύ μεγαλύτερη η δραστηριότητα αυτή. Συνεπώς οι γεωργοί δεν έχουν μεγάλο ειδικό βάρος αν συγκρίνει κανείς την κατάστασή τους με την κατάσταση αυτών οι οποίοι πολλούν τα προϊόντα των αγροτών στον υπόλοιπο κόσμο είτε πολλούν προϊόντα άμεσα στους γεωργούς. Υπάρχει μια διαφορά κλίμακα στο μέγεθος αυτό. Μιλάμε για την αλυσίδα η οποία υποτίθεται λειτουργεί από τον Γεωργό μέχρι το τελικό κατάστημα πώλησης. Τι γίνεται πριν φτάσουμε στο Γεωργό. Θα καταθέσω τροπολογίες λοιπόν οι οποίες θα μας επιτρέψουν να λάβουμε υπόψη μας το τι συμβαίνει πριν φτάσει κανείς στο Γεωργό και τι συμβαίνει φυσικά και μετά. Είμαστε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. και καλό είναι να κάνουμε παρατηρήσεις και να έχουμε αιτήματα σχετικά με την υγεία, την υγιεινή κτλ. Καλά κάνουμε και το κάνουμε γιατί έτσι και αλλιώ η γεωργία παίζει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο περιβάλλον και επηρεάζει άμεσα το περιβάλλον. και η γεωργία και η υλοτομία είναι καθοριστικές για το περιβάλλον. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αμείβουμε σωστά τους γεωργούς για την παραγωγή τους και για προϊόντα τα οποία δυσκολεύονται να διαθέσουν άμεσα οι ίδιοι στην αγορά. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους έτσι ώστε δίκαια οι γεωργοί να φροντίσουν το περιβάλλον και να προστατεύσουν το περιβάλλον, να προστατεύσουν τους υδάτινους πόρους κτλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να πω ότι χαιρετίζω την έκθεση, τη γνωμοδότηση της Έστερ Χαράντς Γκαρσία. Είναι σύντομη, περιεκτική και πολύ εστιασμένη. Συμφωνώ με αυτά που έγραψε. Είναι νομίζω σημαντικό να υπάρξει γνωμοδότηση στην έκθεση Μποβέ. Πολύ συζητήσαμε και στην Επιτροπή Γεωργίας και αλλού στο Κοινοβούλιο για τον τομέα των γαλακτοκομικών ο οποίος στην Ευρώπη είναι πολύ ενδεικτικός και εδώ είναι πολύ σχετική η γνωμοδότηση της κυρίας Γκαρσία. Φαντα... Υποθέτω ότι θα καταλαβαίνουν τα μέλη της Επιτροπής μας ότι όταν επισκεφθείτε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ και αν θέλετε να πάρετε ένα λίτρο γάλα, πάντα βλέπετε ότι το γάλα είναι στα πίσω ράφια του σούπερ Πρέπει να περάσετε όλα τα άλλα ράφια και να δείτε ένα σωρό προϊόντα. Βεβαίως η ελπίδα είναι να γεμίσει το ε, καλαθάκι σας με πολλά άλλα προϊόντα. Γιατί το κάνουν. Ναι, βέβαια παίζει ρόλο ότι είναι ε, βασικό προϊόν. Τώρα πουλιέται στη μισή τιμή του εμφιαλωμένου νερού το γάλα δεν χρειάζεται δηλαδή, ε, δεν χρειάζεται βέβαια ο κτηνίατρος για το προϊόν του, εμφιαλωμένου νερού. Δηλαδή ε, είναι τρελές ε, οι τιμές και πώς εκφράζονται στην τιμή. Οι λιανέμποροι είναι εκείνοι που επιτυγχάνουν τρελά κέρδη σε βάρος των γεωργών, των αγροτών που πληρώνονται λιγότερα από το κόστος παραγωγής για ένα λίτρο γάλα. Εφτά μέρες τη βδομάδα, 365 μέρες το χρόνο χρειάζεται φροντίδα το κοπάδι. Είναι τρομερά κεφαλαιοβόρος ε, ε κλάδος το να έχει κανείς ε, ε, ένα κοπάδι το οποίο και να παράγει γαλακτοκομικά ε, φιλικά προς το περιβάλλον υψηλής ποιότητας. Πώς είναι δυνατόν να επιβιώσουν λοιπόν όταν τους γδέρνουν τα σούπερ μάρκετ, τους αγρότες. Πριν από δύο εβδομάδες ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο ανακάλυψε η κυβέρνηση ότι υπήρχε καρτέλ που λειτουργούσε μεταξύ των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ ούτως ώστε να συμπιέζονται οι τιμές του γάλακτος και όλοι συμφωνούσαν στο καρτέλ να πουλάνε σε πολύ χαμηλές τιμές το γάλα παρά τις επανειλημμένες προσφυγές και από τους αγρότες και από τις ενώσεις τους. Και, και ε, βεβαίως επευλήθησαν ε, πολύ μεγάλα πρόστιμα σε αυτά τα σούπερ μάρκετ. Αλλά αυτά είναι η κορυφή του παγόβουνου. Ξέρω από τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτών ότι ο, ο εισηγητής προτείνει σε όλα τα κράτη-μέλη να θεσμοθετηθεί ένας όμπουτσμεν ο οποίος θα διαιτητεύει μεταξύ ε, αγωγών, ε, σε προσφυγών μεταξύ παραγωγών και λιανεμπόρων. Είμαι υπέρ και γενικά νομίζω ότι και εδώ η γνωμοδότης κυρίας Εράνς Γκαρσία είναι πολύ καλή και ελπίζω να κάνει μια διαφορά, να αλλάξει λίγο τα πράγματα η έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ζωάου Φερέρα. Ευχαριστώ κύριε Σίβενσον. Ευχαριστώ πρόεδρε. <clears throat> θα ήθελα ξεκινώντας να ευχαριστήσω τον εισηγητή, την εισηγήτρια, την κυρία Ερανγκασία. Η γνωμοδότηση περιλαμβάνει καθοριστικές πλευρές του προβλήματος. Ασκείται κριτική στα πλαίσια της ανεπάρκειας των μέτρων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά επίσης ε, ακούγονται και ορισμένα επιχειρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία θα έλεγα, στα οποία ασκείται κριτική ακούγεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στην υψηλή τιμή την οποία πληρώνει ο καταναλωτής με τη χαμηλή τιμή την οποία πληρώνεται ο γεωργός. Δεν είναι δυνατό να υποστηρίζουμε τέτοιες απόψεις και έτσι για αλλιώς είμαστε υποχρεωμένοι να προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε τις πιο ευάλωτες, τα πιο ευάλωτα τμήματα αυτής της αλυσίδας. <clears throat> Όσο όμως αναποτελεσματικές είναι αρχές επί του προϋπολογισμού, ασκούνται πάρα πολλές, ε, θα έλεγα, καταχρηστικές μέθοδοι οι οποίες ευνοούν τον μεταποιητή, ευνοούν τον έμπορο και δημιουργούν αρνητικά για τον γεωργό. Συνεπώς, θα πρέπει να ξεπεράσουμε νομίζω κάποια από τα πλαίσια τα οποία θέτει η κυρία Έραντς. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις πραγματικές αιτίες του προβλήματος, τι μας έχει οδηγήσει στις αιτίες αυτές μάλλον. Και να, ε, τότε μόνο να μπορέσουμε να αναζητήσουμε τις πραγματικές λύσεις. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε σαν παράδειγμα να δούμε τι συνέπειες προκαλεί για την ύπεθρο χώρα η απώλεια εισοδήματος των γεωργών. Πολύ συχνά μιλάμε για την ασφάλεια των τροφίμων και το περιβάλλον στην Επιτροπή μας και ταυτόχρονα διαπιστώνουμε την εγκατάλειψη διαφόρων μορφής παραγωγής στην ύπεθρο της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Έχουν εγκαταληφθεί βέβαια σε ορισμένες χώρες και κάποια εκτατικά συστήματα καλλιέργειας τα οποία είναι ασύμβατα με την προστασία της ε, <clears throat> βιοπικιλότητας. Βλέπουμε λοιπόν ότι ταυτόχρονα με την εγκατάλειψη αυτών των μορφών παραγωγής σε ορισμένες περιοχές υιοθετούνται σε άλλες περιοχές. Συνεπώς ολόκληρες περιφέρειες σήμερα χαρακτηρίζονται από μια υπερβολική έκθεση σε φυσικές καταστροφές γιατί κανένας δεν τις κατοικεί. Υπάρχει και η εντατικοποίηση της παραγωγής σε συγκεκριμένες περιφέρειες με ό,τι συνέπειες αυτό προκαλεί στο περιβάλλον. Υπάρχει επίσης και αύξηση της εξάρτησης της ε, τροφιμικής από άλλες χώρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις η εξάρτηση αυτή φτάνει το 75% κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Δεν θα ήθελα να απαριθμίσω όλα τα προβλήματα. Οι συνάδελφοι το έκαναν αυτό και σωστά έκαναν. Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να δούμε ποιες είναι οι αιτίες των προβλημάτων. Και να πούμε ότι πολλά από τα προβλήματα αυτά είναι συνέπειες της κοινή αγροτικής πολιτικής όπως υπάρχει σήμερα. Απελευθερώθηκε πλήρως η αγορά των γεωργικών προϊόντων. Η προστασία της γεωργικής παραγωγής είναι ανεπαρκεστάτη. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Η παραγωγή τροφίμων από μόνη της έχει πάρα πολύ μεγάλη ουσία και δεν θα πρέπει να υπόκειται στις διακυμάνσεις της αγοράς και στα καπρίτσια της αγοράς. Η απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου θα πρέπει επίσης να μην ασκεί τέτοιου είδους πιέσεις προς τις τιμές. Τιμές οι οποίες πληρώνονται στον καταναλωτή, αλλά από τον καταναλωτή, αλλά και τιμές οι οποίες πληρώνονται στον παραγωγό και οι οποίες πολλές φορές είναι ιδιαίτερα χαμηλές. Σε επίπεδο λοιπόν θεσμικό και σε επίπεδο νομοθετικό, στην ουσία έχουμε λόγω ακριβώς αυτού του επίπεδου πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς, έχουμε ανοίξει τις πύλες σε καταχρήσεις από όλες τις πλευρές. Τίθενται λοιπόν δύο βασικές ερωτήσεις στα πλαίσια της γνωμοδότησης Έραντς Γκαρσία. Πρώτον, το θέμα της ρύθμισης της αγοράς. Και δεύτερον, ο καθορισμός σωστών τιμών για τους παραγωγούς. και συμπληρωματικά τίθεται επίσης και το θέμα των κοινοτικών προτιμήσεων. Ξέρουμε ότι υπάρχουν εισαγωγές από τρίτες χώρες. Οι εισαγωγές αυτές θα πρέπει να βασίζονται στην αρχή της συμπληρωματικότητας και όχι σε αυστηρά εμπορικές αρχές και σε μια λογική ανταγωνιστική επίσης. Αυτά τα είπαν άλλωστε και οι προλαλήσαντες συνάδελφοι για λόγους διασφάλισης των προμηθειών σε τρόφιμα θα πρέπει να λάβουμε μέτρα, αλλά μην ξεχνάμε και άλλους λόγους, κοινωνικούς λόγους, περιβαλλοντικούς λόγους, αποκατάσταση του κοινωνικού ιστού που έχει τροφή σε συγκεκριμένες περιοχές της υπαίθρου αγροτικές κτλ. Η γνωμοδότηση λοιπόν που έχουμε μπροστά μας λέγει ότι δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στις ε, τιμές τις υψηλές που πληρώνει ο καταναλωτής και στις χαμηλές τιμές με τις οποίες πληρώνεται ο παραγωγός. Αυτό δεν είναι λογικό. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε με ποιο τρόπο σχετίζονται οι δύο αυτές τιμές. Και θα πρέπει να υπάρχουν κάποια περιθώρια εμπορίας των γεωργικών προϊόντων ευρύτατα. Αυτό θα ήταν ένα μέσο το οποίο ουσιαστικά θα δημιουργήσει ένα ανώτατο, μία ανώτατη τιμή αν θέλετε και έτσι θα έχουμε μία ικανοποιητική τιμή που να πληρώνεται στον παραγωγό και μία ικανοποιητική τιμή ε, που θα πληρώνει ο καταναλωτής. Μείωση δηλαδή ουσιαστικά του περιθωρίου κέρδους των ενδιαμέσων σταδίων. Αυτό είναι ένα επιπλέον σημείο το οποίο θα πρέπει να προσθεθεί στην γνωμοδότηση. Λοιπόν, δίκαιες τιμές για τους γεωργούς, για τους παραγωγούς, έτσι ώστε να μην εγκαταλείψουν τις δραστηριότητες παραγωγής τους. Σας ευχαριστώ. Κύριε Γκροστέτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στη γνωμοδότηση της κυρίας Εράνς υπάρχουν στοιχεία ουσιώδους σημασίας για τη μελλοντική ε, γεωργική πολιτική. Γιατί είναι ουσιαστικά αυτά, γιατί ζητάμε όλο και περισσότερα από τους αγρότες να εξασφαλίζουν την επιστημιστική σταθερότητα και ασφάλεια στην Ευρώπη, είναι σημαντικό. Τους ζητάμε περισσότερα περιβαλλοντικά πρότυπα και με ασφάλεια να παράγουν τρόφιμα για τους καταναλωτές και ταυτόχρονα που τους τα ζητάμε όλα αυτά συμμετέχουν και στη χωροταξία οι αγρότες. Δηλαδή, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε γεωργούς στην Ευρώπη, αγρότες, και θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Έτσι ώστε αυτά που ζουν σήμερα οι αγρότες μας να μην συνεχιστούν, ε, πέφτουν συνέχεια τιμές των ε, πρώτων υλών δηλαδή τη τιμές παραγωγού στα τρόφιμα και θα πρέπει να τη σταματήσουμε, να τη ρυθμίσουμε αυτή τη μείωση και να καταπολεμήσουμε ε, την πτητικότητα των τιμών των γεωργικών προϊόντων. Είναι πολύ σημαντική γνωμοδότηση για μένα, θα σας αναφέρω δύο μόνο στοιχεία. Πρώτον, θεωρώ σημαντικό να ρυθμίσουμε το θέμα της κατανομής της προστιθέμενης αξίας στη διατροφική αλυσίδα και ε, της διαπραγματεύσεις παραγωγών με διανομής. Εδώ μπαίνει ένα ζήτημα ενίσχυσης των οργανώσεων παραγωγών και είναι γεγονός ότι έχουμε μια σύγκρουση μεταξύ του ευρωπαϊκού δικαίου ανταγωνισμού και ε, των ε, γεωργικών επαγγελμάτων. συστηματικές συμβάσεις. Πολύ σημαντικό. Να έχουμε μια στοιχειώδη ρύθμιση, εν πάση περιπτώσει, τη κοινή γεωργική πολιτική. Επιτρέψτε μου να φέρω και ένα άλλο πρόβλημα, που είναι η αφανή ε, φορεί ε, τη τροφική αλυσίδα. Για παράδειγμα, όταν είχαμε την κρίση στο γάλα, θεωρήσαμε ότι αυτό οφειλόταν στη μαζική εισαγωγή φθηνού γάλακτος από τη μεγάλη διανομή και τη βιομηχανία τύπου Nestlé, και τα λοιπά, μεγάλες εταιρείες. Όμως έγινε μια μελέτη μετά ε, στα τελωνία και διαπιστώσαμε ότι το γάλα εισήχθη κυρίως από οργανισμούς ε, συλλογικής σύτησης, σοντεξό και τα λοιπά, που κάθε μέρα ε, δίνουν ένα εκατομμύριο μερίδες ή ε, κάποιες εταιρείες τύπου William Seran και τα λοιπά που ε, παράγουν και πουλάνε έτοιμες μερίδες φαγητού. Αυτοί λοιπόν διατάραξαν και οδήγησαν σε προβλήματα στην τιμή του γάλακτο στην αγορά και όχι μεγάλες εταιρείες. 20% ε, των ε, μερίδων ε, που παρασκευάζονται καλύπτονται από προϊόντα εισαγόμενα και όταν μιλάμε για τη διατροφική αλυσίδα πολύ συχνά ξεχνάμε αυτούς τους αθέατους φορείς της αγοράς. Είναι μια μεταβιοποιητική μεταποιητική συγγνώμη βιομηχανία αυτή που δεν λαμβάνεται υπόψη δεν είναι παραγωγή τροφίμων, είναι παραγωγή τίμων φαγητών και ε, ασκούν αθέμητο ανταγωνισμό στην κλασική διατροφική αλυσίδα. Θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό για να βοηθήσουμε τους αγρότες μας για να είναι αρκετά ισχυροί απέναντι σε αυτές τις πρακτικές. Διότι τελικά αυτές διαταράσσουν απολύτως την αγορά σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Γκροστέτη, κυρία Κλάσσα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τώρα, ε, όλοι έθεσαν το ερώτημα τι θα κάνει η Επιτροπή μας ε, για το θέμα αυτό των αγροτών και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ε, αλυσίδα εφοδιασμού στην Ευρώπη. Μπορούμε και στη Γεωργική Επιτροπή, υπάρχει η Επιτροπή της Εσωτερικής Αγοράς. Όμως έδειξε η συζήτηση ότι πολύ σωστά κάνουμε και ασχολούμεθα υπεύθυνα με το θέμα αυτό τις τιμές υγιεινών τροφίμων γιατί τα προϊόντα αυτά που πολύ σωστά τα ε, συνοδεύουμε με προϋποθέσεις, προδιαγραφές, όρους για υγιεινή, καλό περιβάλλον, ποιότητα. Ε, τέτοια προϊόντα πρέπει να φτάνουν στην αγορά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να ενδιαφερόμαστε και για την αγορά και το μερίδιο που έχουν αυτά τα προϊόντα. Θέλω να υπογραμμίσω άλλη μια φορά ότι πρέπει να είναι δυνατόν να υπάρχει ανταποδοτικότητα στο σύστημα και να υπάρχει δυνατότητα να αμείβεται ε, σωστά ο αγρότης μέσα από την αγορά. Δεν μπορεί ένα ψωμάκι να ε, για ένα ψωμάκι να παίρνει δύο σέντο αγρότης μόνο για το ε, αλεύρι που έβαλε, είναι πάρα πολύ χαμηλό το κόστος. Πόσο συγκεκριμένη μπορεί να είναι μια τέτοια γνωμοδότηση και ποιο είναι το όριο μεταξύ ρύθμισης της αγοράς πολύ αυστηρής και μιας κοινωνικής οικονομίας της αγοράς που αφήνει και ελευθερία. Υπάρχει μια διαφορά. Θέλω να ευχαριστήσω τη συνάδελφο γιατί αφενός δεν είναι εδώ. Όχι, εδώ είναι. Κατάφερε αφενός σε έξι σημεία να συνοψίσει τα βασικά, να παριθμίσει τα σημαντικά. Στο σημείο έξι ε, θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, γιατί ανοίγει ένα πολύ σημαντικό θέμα. Λέει, μιλάει για καλύτερη ενσωμάτωση των διαφόρων κρίκων της αλυσίδα σε διαπαγγελματικέ οργανώσεις και μιλάει για κωδιδίκες ορθών πρακτικών, τυποποιημένες εθελοντικές συμβάσεις. Το ερώτημα είναι, αρκούν οι τυποποιημένες εθελοντικές συμβάσεις ή μήπως χρειάζεται κάτι παραπάνω. Κάποιος μηχανισμός της αγορά ιδιαίτερα για τις διεπαγγελματικές οργανώσει, ούτως ώστε όταν πρόκειται ας πούμε για ευαλείωτα προϊόντα, φρέσκα, ε, με βιταμίνες, ε, ε, προκυπευτικά κλπ. Ε, για αυτά τα προϊόντα να βρούμε καινούριου πιο ευέλικτους κανόνες και ρυθμίσεις που θα είναι διαφορετικές από ένα προϊόν που έχει μακρύ κύκλο ζωής στο ράφι. Χρειάζονται επίσης ε, συζητήσεις και συντονισμός για τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τιμές. Θα πρέπει να τα παρακολουθούμε από κοντά όλα αυτά γιατί είναι σημαντικός ο στόχος εδώ. Πώς θα μπορέσουν τα καλά προϊόντα που ανταποκρίνονται σε όλες τις ε, σωστές προδιαγραφές, πώς θα φτάσουν να πολλούνται περισσότερα στην αγορά, προάγοντας έτσι την κουλτούρα μας ε, για το περιβάλλον, το την υγιεινή των τροφίμων και την ύπεθρο. Η κυρία γνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται ένα σούπερ μάρκετ λέει πάρα πολλά από τον τρόπο και την οτροπία με τον οποίο οργανώνεται μια χώρα. Σαν παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο ο κόσμος τσακώνεται με τα έτοιμα φαγητά πριν φτάσει στο γάλα. Σε ένα Ολλανδικό βέβαια σούπερ μάρκετ οι άνθρωποι τρέχουν πρώτα στα γαλακτοκομικά προϊόντα αλλά και προέρχομαι από γαλακτοπαραγωγό περιοχή και αυτό είναι φυσιολογικό. Και τώρα στα Ολλανδικά σοβαρά για τη γνωμοδότηση. Πολλοί συνάδελφοι μίλησαν και τους ευχαριστώ. Είναι όντως σημαντικό το θέμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά την κυρία Εράντς ε, για την γνωμοδότηση της που είναι και καλή και συνεκτική και σύντομη. Ε, είναι και μέλος στην Επιτροπή Γεωργίας η κυρία Εράντς και βέβαια γνωρίζει ε, μέχρι τελευταία σκεραία το θέμα και η δική μου πρώτη αντίδραση ήταν «Μα δουλειά έχουμε τώρα εμείς ε, ως Επιτροπή Περιβάλλοντος. Πρέπει να κάνουμε ξεχωριστή γνωμοδότηση. Είναι θέμα τη γεωργίας. Ε, και είναι θέμα ανταγωνισμού, ε, είναι θέμα όμως και βιομηχανίας και καταναλωτών. Καμιά φορά το ξεχνάμε ότι η έκθεση έχει να κάνει και με τους καταναλωτές και ότι τα κέρδη δεν κατανέμονται δίκαια ε, στη διατροφική αλυσίδα και ο αγρότης δεν παίρνει σχεδόν τίποτα. Λοιπόν, δεν είναι θέμα γεωργίας, υπάρχει και σκοπιά του καταναλωτή. Και αν δείτε τις τιμές καταναλωτού και τις τιμές ε, παραγωγού και πώς ανοίγει η ψαλίδα, τότε είναι θέμα ακριβώς που πρέπει να, ε, να εξεταστεί όταν ε, τα σιτηρά αυξάνονται, αυξάνεται και το ψωμί. Όταν μειώνεται τα σιτηρά, δεν μειώνεται το ψωμί. Γι' αυτό ανοίγει αυτή η ψαλίδα και έρχεται και ο καταναλωτής στη μέση να διαμαρτυρηθεί. Και εγώ δεν λέω να αυξηθεί η τιμή ε, καταναλωτού, αλλά να υπάρχει μια σωστή κατανομή των κερδών. Αλλά παρακαλώ προσέξτε με τη γνωμοδότηση αυτή να μην κάνουμε συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής γεωργίας και να μην βάζει ο καθένας ό,τι θέλει για τη μελλοντική γεωργία. Πολύ καλά τα λέτε και τα σκέφτεστε, αλλά δεν είναι του παρόντος. Ποιο είναι το πρόβλημα και ο πυρήνα του άνδρου, το θέμα που μας απασχολεί εμάς, που είναι το περιβάλλον και η δημόσια υγεία. Στο περιβάλλον το πρόβλημα είναι το εξή. Το είπε και η κυρία Γκροστέτ προηγουμένω. Για του παραγωγού. τους ζητάμε και περιμένουμε να κάνουν διάφορα για τη βιοπικιλότητα, για το τοπίο, για τη διατήρηση του περιβάλλοντος και μια σειρά άλλα πράγματα. Και από την άλλη ο, ο παραγωγός που είναι η πρωτογενής ε, παραγωγή ε, είναι εκείνος που πληρώνει τα σπασμένα στις τιμές. Τα μοιράζονται όλοι οι υπόλοιποι τα κέρδη και ό,τι περισσεύει πάει στον παραγωγό και στον αγρότη. Και στη δική μου χώρα δεν αρκεί αυτό παρόλο που η χώρα μου είναι πολύ γεωργική, συχνά δεν αρκούν αυτά τα χρήματα για να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπέ εισόδημα σε ένα αγρότη. Για να μην μιλήσω ε, καν για τις υπόλοιπες δραστηριότητε που απαιτούμε από τον αγρότη. Περιβάλλον, βιοπικιλότητα, υγιεινή κτλ. Φροντίδα του τοπίου. Λοιπόν, θα πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό αν θέλουμε διαφορετική πολιτική γεωργία, αν θέλουμε να ανταμείβουμε και να επιβραβεύουμε και να πληρώνουμε του αγρότε για όλα αυτά που του ζητάμε να κάνουν εκτό από την παραγωγή, ε, τότε κάπω θα πρέπει να βάλουμε το χέρι στην τσέπη. Δεν ξέρω αν αυτό είναι επιδοτήσει ή πιο σωστή τιμή των προϊόντων, θα το ξανασυζητήσουμε. Για τη δημόσια υγεία, συμφωνώ, Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη. Η ασφάλεια των τροφίμων και επιστηστική ασφάλεια να έχουμε αρκετά τρόφιμα, γιατί ένας αγρότης που εγκαταλείπει την εκμετάλλευση δεν θα πάει να ξαναγίνει αγρότης. Στη χώρα μου που υπάρχει πρόβλημα στέγης και ψάχνουμε το κάθε τετραγωνικό εκατοστό, μόλις ένα αγρόκτημα σταματήσει τη λειτουργία του γίνεται αμέσω κατοικία. Και ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν ε, να διατηρήσουμε και τους αγρότες στην ε, Ήπεθρο και να έχει ένα αξιοπρεπές εισόδημα για την παραγωγή ο αγρότης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Εράνς. Πραγματικά έχει κάνει πολύ καλή προσπάθεια. Θα κάνω και εγώ κάποιες τροπολογίες. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, Esther Hader. Ευχαριστώ, Γιάννος Χάντερ. Κυρία Πρόεδρε, ακούγοντας ε, τη συζήτηση, σχολιάζω τα εξής ίσως ό,τι αφορά τα θέματα αρμοδιότητας κομισιών γιατί το πρώτο θέμα είναι η ασφάλεια των τροφίμων έχω την εντύπωση βλέποντας την, τις ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι δεν ξέρει δεξιά τι πει η αριστερά. Δηλαδή, αφενός έχουμε πολύ αυστηρές διατάξεις για την ασφάλεια των τροφίμων που πρέπει να εφαρμόζονται και οι Πολωνοί και οι Ούγγροι και οι Γάλλοι και όλοι τέλο πάντων ενώ από την άλλη πλευρά στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχονται και τρόφιμα που δεν ανταποκρίνονται καθόλου και δεν πληρούν καθόλου τις αυστηρές προδιαγραφές στην Ουγγαρία. Πρόσφατα είδαμε πολλά σκάνδαλα, θα σας πω δύο. Είχαμε ε, πουλερικά με διοξίνες που πέρασαν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έφτασαν και σε εμά, όπως επίσης και ξηρούς καρπούς με αφλατοξίνες από το Μαρόκο. Και στις δύο περιπτώσεις είχαμε ε, οριακές τιμές που ξεπερνούσαν, μάλλον όχι, ε, διαπιστώθηκαν τιμές που ξεπερνούσαν κατά πολύ τις ε, οριακές. Και αναρωτιέμαι, τα κάνουμε σωστά. Γιατί είναι σαφές ότι εδώ θα πρέπει να γίνουμε πολύ πιο αυστηροί, να δείξουμε πολύ μεγαλύτερη συνέπεια για να προστατέψουμε την αγορά μας και τα τρόφιμά μας, για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας και την δική μας κατανάλωση των τροφίμων. Είναι σημαντικό αυτό και για τους αγρότες μας. και για τα προϊόντα που έρχονται σε εμά από τρίτες χώρες. Λοιπόν, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Από τη μια είμαστε αυστηρότατοι και από την άλλη ε, τρώμε και ε, καθόλου ασφαλή προϊόντα καμιά φορά. Τώρα, στην έκθεση λέει επίσης ότι, για παράδειγμα, πρέπει να περιορίσουμε τα μονοπόλια στην αγορά. Και ε, εδώ θα σας πω ένα παράδειγμα από τη χώρα μου, την Ουγγαρία. Καμιά φορά πέφτουν οι τιμές για κάποιους λόγους συγκεκριμένους. Στην Ουγγαρία υπάρχουν 96 νομικές βάσεις για τη μείωση των τιμών. Δηλαδή παίρνουν 20 με 25% κάτω της καθορισμένης τιμής για τον καταναλωτή. Και αυτό δεν το βλέπουμε μόνο στην Ουγγαρία αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτή είναι μια κατάχρηση της θέσης στην αγορά. Αυτές οι καταχρηστικές πρακτικές ε, θα πρέπει, γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν όχι μόνο στην Ουγγαρία αλλά και αλλού. Και είμαι υπέρ. Ευχαριστώ. η κυρία Καρίνα Φαν Μίκελσον από την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή. Εκτιμώ πολύ το ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για, το, για την τροφική αλυσίδα και τη λειτουργία της και την ε, δίκαιη διανομή. Προσβλέπουμε στη γνωμοδότηση που ετοιμάζεται και θεωρούμε ότι ε, η έκθεση Μποβέ έχει σχέση με την ανακοίνωση και ευθυγραμμίζεται με την ανακοίνωση της Κομισιόν του Νοεμβρίου και του Μαρτίου τα συμπεράσματα του Συμβουλίου φέτος. Στην Κομισιόν μέχρι τον Νοέμβριο αυτού του έτους θα ε, θεσπίσουμε, θα συντάξουμε έκθεση συνέχεια της ανακοίνωσης του φθινοπόρου και επίσης θέλουμε να δημιουργηθεί ένα φόρουμ, αυτό είναι συνέχεια της ομάδας υψηλού επίπεδου για την ανταγωνιστικότητα του ε, τομέα ε, γεωργίας και τροφίμων και θέλουμε να έχουμε ευρεία βάση ε, συμμετοχής από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας για το θέμα και θα περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την τελική έκθεση. Ευχαριστώ. Euh, ε, κυρία Γκαρσία, και σας ευχαριστούμε όλοι γιατί η γνωμοδότησή σας ε, βρήκε ομόφωνη ε, θετική υποδοχή. <laughs> Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Ήταν πολύ επικοδομητικά αυτά που μας είπαν θεωρούν όλοι αναφέρονται στα έξι σημεία, βλέπετε ότι είναι πολύ ε, σύντομη η γνωμοδότηση, πάρα πολύ περιεκτική, ε, μονοσέλιδη. Και θα καταλάβατε ότι επίτηδες έχω κάνει αυτή την προσπάθεια να περιοριστώ σε μία σελίδα. Αν ήθελα να επεκταθώ θα μπορούσα να δώσω και παραδείγματα για κάθε ε, σημείο και θα ήταν πολύ μακροσκελής η έκθεση, αλλά δεν πρόκειται περί αυτού. Αυτό που θέλουμε να στείλουμε σαφέ μήνυμα στην καθήλυνα αρμόδια επιτροπή που είναι η Επιτροπή Γεωργίας να εργαστεί προς την κατεύθυνση αυτή. Και όταν φτάσουμε στην Ολομέλεια, ε, να το ψηφίσουμε στο Στρασβούργο, θα πρέπει όλοι οι παράγοντες αλυσίδας ε, από τον ε, αγρότη, τον παραγωγό μέχρι ε, τον καταναλωτή να καταλάβουν ότι το κοινοβούλιο είναι στο πλευρό του πολίτη. Δεν θέλει καταχρήσει. Οι μικροί παραγωγοί να έχουν τι ίδιε δυνατότητε να ορθοποδούν με τι μεγάλε εταιρείε. Γι' αυτό που μας ενδιαφέρει οι καταναλωτές να έχουν ευρωπαϊκά προϊόντα και εκείνοι που ζουν στην Ήπεθρο να εξακολουθούν να ζουν στην Ήπεθρο και να εργάζονται στη γεωργία ή την κτηνοτροφία και να έχουν εισόδημα. Εμείς δεν θέλουμε να δώσουμε κανένα μετάλλιο στον εαυτό μας παράσημο, τι ωραία έκθεση που κάναμε και τι πολλά λόγια που τα λέμε ωραία. Αυτό που θέλουμε είναι να δώσουμε ένα μήνυμα που να συνοδεύει την Επιτροπή Γεωργίας στην Ολομέλεια. Περιμένω τις τροπολογίες σας και εγώ θα μπορούσα να κάνω τροπολογία ενδεχομένω. Ε, αν θέλετε και μαζί σας μπορούμε να τα ξανακοιτάξουμε ε, θέματα που ενδιαφέρεστε να καταθέσουμε και καμιά κοινή τροπολογία. Πάντως αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως τώρα είναι να δώσουμε ε, εικόνα ενότητας. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ευχαριστώ. Ενθυμίζω ότι η προθεσμία είναι η 10η Μαΐου. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος 2-3 Ιουνίου, στη Γεωργία 28 Ιουνίου και στην Ολομέλεια το Σεπτέμβριο. Τερματίζεται εδώ η συνεδρία μας. Συνεδρίασή μας θα βρεθούμε αύριο στις 9 για τις ψηφοφορίες.